Καλώς ορίσατε στη συνεδρίασή μας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχετε σχόλια, υιοθετείτε η ημερήσια διάταξη, εγκρίνεται, πρέπει να εγκρίνουμε και τα πρακτικά διαφόρων συνεδριάσεων. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνονται τα πρακτικά Έχουμε επίσης μερικές αγγελίες σύμφωνα με τον κανονισμό μας ε, συστάσεις των συντονιστών μετά την ε, συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου για τον διορισμό ε, σχετικά με τα ότιση παράγωγα βάσει των συστάσεων της Κεντρικής Τράπεζας ε, της χορηγήσεις ε, για την ΕΛΚ, αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για την φυρολογία σχετικά ε, με τις διάφορες διαφετήσεις διασυνοριακές. Επίσης στην ΑΛΔΕ το, το φάκελο για τις διασυνοριακές συντάξεις επίσης αντιδράσεις στις συστάσεις σχετικά με την ε, φορολογική αντιμετώπιση στην ΑΛΔΕ, εναρμόνιση της ε, φορολογικής ε, επιβάρυνσης σχετικά με τις, τα πρόστιμα στις τράπεζες εδώ ένα, μια ταχύρυθμη οδός η προθεσμία θα είναι 4 Σεπτεμβρίου για τις ε, τροπολογίες με 25 ε, Σεπτεμβρίου εξέταση των τροπολογιών, επίσης παράλληλες ε, παρουσιάσεις για το τραπεζικό πακέτο ή το χρονοδιάγραμμα θα αναθεωρηθεί εν ευθέτω χρόνο εφόσον θα ψηφίσουμε και αύριο σήμερα για την πρώτη παρουσίαση σχετικά με τις, τα μεγάλα ανοίγματα. Οι συντονιστές αποφάσισαν να αναβάλουν για το 2018 την αποστολή στο Μπεϊτζίν και στη Σανγκάη. Αποφασίστηκε να ζητήσουμε άδεια για έναν πρόσθετο προορισμό ε, τον Οκτώβριο για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και 2 και 3 ε, Νοεμβρίου στην Πορτογαλία, εάν υπάρχουν βεβαίως διαθέσιμοι συνομιλητές. Επίσης, 22 ε, Σεπτεμβρίου δεν θα λάβει χώρα η συνεδρία των κοσμητόρων για ε, τις εξουσιοδιοτημένες πράξεις, επίσης την κακή πώληση των προϊόντων που ήταν αντικείμενο αναφορών, οι συντονιστές αποφάσισαν για τις απαντήσεις σχετικά με την αναφορά 0709 3, 5, 79, 2016 σχετικά με τις ε, ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις. Με συγχωρείτε για αυτόν την ε, φόρτο εργασίας που έχουμε πριν από τον διάλογο. 28 Ιουνίου οι Επιτροπές Λίμπε και ΕΚΟΝ είχαν την τελευταία τους συνεδρίαση ε, με ε, Προεδρία Μάλτας σχετικά. Το μόνο θέμα ήταν η δημόσια πρόσβαση για Προεδρία της Μάλτας πέριξε για τα τράστα αυτά δεν έχει για τα καταπιστεύματα αυτά δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Ε, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με τριμερή διάλογο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Εστονίας και θα λάβει χώρα αύριο. Ο τριμερής αυτός διάλογος. FSI. Έγινε κάποια πρόεδρος μετά τον τριμερή διάλογο της 21 Ιουνίου ε, για την αναθεώρηση του κανονισμού ΕΦΣΑ για προπαραγωγική συζήτηση για θέματα σχετικά με την ανώτατη οροφή και για την υπαγωγή και τα scoreboard. Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν μετά σε τεχνικό επίπεδο για ε, για κάποια εναρμόνιση και όλα τα μέρη μπόρεσαν να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για τα περισσότερα πολιτικά θέματα, ε, άλλα θέματα για συζήτηση, κυρίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση, διακυβέρνηση, φορολόγηση και ο επόμενος διάλογος ο τριμερής θα λάβει χώρα αύριο επίσης. Και τώρα τέλος, με χαρά, θα ήθελα να καλωσορίσω σήμερα τον καθηγητή Νίλ Στίγκεσεν, που είναι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Να τον ευχαριστήσω διότι δέχτηκε ε, με χαρά την ε, πρόσκλησή μας ε, να έρθει εδώ για ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής. Είχαμε ήδη μια ανταλλαγή απόψεων τον Δεκέμβριο με τον καθηγητή Τίγκεσαν μετά το διορισμό του και αποφάσισε να έρθει σε τακτική συνεδρίαση για να μας μιλήσει για την ε, δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου ε, σχετικά με το εξάμεινο. Ο καθηγητής Στίγκισον ε, συμμετείχε στην συνεδρίαση του Eurogroup και το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο δημοσίευσε μια έκθεση για τις προπτικές του δημοσιονομικού προσανατολισμού, του fiscal stance και θα θέλαμε την αξιολόγησή σας και τα ε, συμπεράσματα. Ε, εγώ ε, έτεινα να υποστηρίξω την Επιτροπή, αλλά η έκθεση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και καλύπτει πάρα πολλά προβλήματα και θέματα. Υπάρχει έλλειψη συντονισμού, αν κάποιος θέλει να έχει μια μια πλήρη συντονισμένη θέση σχετικά με τον δημοσιονομικό αυτόν προσανατολισμό. Δεν έχουμε βεβαίω τα εργαλεία για αυτό το θέμα. Απ' την άλλη πλευρά, αν θέλουμε ένα δημοσιονομικό προσανατολισμό που να βασίζεται σε καλή αξιολόγηση της κατάστασης σε κάθε χώρα, διότι έχουμε ε, χώρες ε, που έχουν μικρότερο ή μεγαλύτερο προσανατολισμό ε, και έχουν τότε ορισμένα περιορισμούς πρακτικούς και νομικούς. Βεβαίως μετά την παρουσίασή σας θα μπορέσουμε και η Κομισιόν θέλει να βεβαίως να έχει ορισμένα ποσοτικές εκτιμήσεις. Βεβαίως η μήτρα αυτή δεν αναθεωρήθηκε και από την άλλη πλευρά η Κομισιόν θα κάνει τις κατάλληλες εκτιμήσεις για κάθε χώρα για τις διαρθρωτικές προσαρμογές που απαιτούνται από τη Μήτρα. Και για να κάνουμε μια διάκριση νομική ανάμεσα στις διατάξεις, στις δημοσιονομικές που απαιτούνται από την εφαρμογή και ποιο είναι το περιθώριο εκτίμησης από την Κομισιό ε, για να έχουμε ε, βάση των συνεπειών της ατελούς εφαρμογής του κανόνα. Και ελπίζω ότι θα βεβαίως θα οδηγηθούμε σε μια λύση του διλήμματος όπου έχουμε. Θα ακούσουμε όμως πρώτα τις απόψεις για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι που βρίσκεστε εδώ και έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Κουαλτιέρη και μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Πράγματι είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ. Εκτιμώ την πρόσκλησή σας. Τον προηγούμενο Δεκέμβριο είχα μια σύντομη βιντεοδιάσκεψη με κάποια μέλη της Επιτροπής σας ε, και είναι επίσης κάτι που εκτίμησα. Ε, συμμετείχα στο ακαδημαϊκό πάνελ ε, για την προετοιμασία της ε, ακρόασης του διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, πάντα εκτιμούσα τη δουλειά που κάνετε στον τομέα της οικονομικής πολιτικής ε, και άλλους τομείς. Βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω την ε, πρώτη έκθεση που έχουμε εκπονήσει στο Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Διοριστήκαμε πέρσι τον Οκτώβριο και πλήρη γραμματεία είχαμε πλέον από την 1η Μαρτίου. Ο Μάρτιν Λάρτς που βρίσκεται δίπλα μου είναι ο επικεφαλής της γραμματείας μας. Η πρώτη μας έκθεση είναι σχετικά σύντομη και ελπίζω σχετικά ευανάγνωστη. Καταρχάς επικεντρωθήκαμε στη, στο δημοσιονομικό προσανατολισμό για την ε, περιοχή του ευρώ για το χώρο του ευρώ στο σύνολό της. Και η προσέγγιση σχετίζεται με την εντολή μας. Εξετάσαμε λοιπόν το δημοσιονομικό προσανατολισμό με βάση ε, την ε, οικονομική εκτίμηση και αυτό μάλιστα είναι το πρώτο τμήμα της εντολής μας. Επικεντρωνόμαστε στο έτος 2018 και εξετάζουμε αναλυτικά τις εθνικές πολιτικές επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με, την, με το δημοσιονομικό προσανατολισμό της Ευρωζώνης ε, λόγω του πόσο επίκαιρο είναι το θέμα αυτό. Συζητήθηκε ε, εντατικά και πέρσι και στην Ευρώπη και αλλού και αποτελεί τη μία πτυχή της εντολής μας. Η άλλη είναι <clears throat> η εφαρμογή των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων γιατί επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με τον δημοσιονομικό προσανατολισμό. Αυτό συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Την Άνοιξη θα πρέπει να υποβάλουμε συστάσεις ε, για την Ευρωζώνη και ε, για να βοηθήσουμε να στην προετοιμασία των προϋπολογισμών το φθινόπωρο και γι' αυτό ήταν φυσική ακολουθία για μας να ξεκινήσουμε από αυτό και κατόπιν να προχωρήσουμε στις πιο αναλυτικές εργασίες σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών κανόνων ε, και άλλες πτυχές που αναφέρετε εσείς στην εισαγωγή σας. Στο πλαίσιο αυτού του εγχειρήματο ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε και τη βοήθεια των ε, εθνικών ε, δημοσιονομικών συμβουλίων των χωρών με τις οποίες θα ασχοληθούμε. Προσπαθούμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση στην Ευρωζώνη με βάση μια σειρά προβλέψεων και αναλύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του ΟΣΑ, του Δουνουτού και ιδιωτικών φορέων. Καταλαβαίνουμε επίσης ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο σε μία σειρά δικτών, δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να ασχοληθούμε μόνο με, την, ε, με το χάσμα στην παραγωγή. Θα πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα ε, γιατί αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο θα έχουμε αύξηση των τιμών και θα δούμε τελικά πλεόνασμα σε κάποιους τομείς. Ε, όταν εφωνήθηκε η συνθήκη του Μάστριχτ, ε, μίλησαν κάποιοι κατά της ε, αναλυτικής ρύθμισης ε, όσον αφορά το δημοσιονομικό προσανατολισμό. Εμείς λοιπόν δεν προτείνουμε ούτε και εμείς αυτό το fiscal fine-tuning. Δεν πιστεύουμε ότι δικαιολογείται κάτι τέτοιο. Ενδιαφέρον είναι το αν αυτό που προτείνουμε ε, συμμορφώνεται με τους δημοσιονομικούς κανόνες ε, και μπορεί να εφαρμοστεί δημοσιονομικό προσανατολισμό ε, στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση, η συνένεση σε όλε τι πηγέ που σα ανέφερα είναι ότι ότι αποκαθίσταται η οικονομία, αλλά απομένουν πολλά να γίνουν ακόμα, διότι υπάρχει ανεργία, υπάρχει ε, ανεπαρκής, υπάρχουν ανεπαρκείς επενδύσεις ε, και ήδη αναφέρθηκα στο πλεόνασμα του ισολογισμού. Ακόμα η οικονομική πολιτική είναι ιδιαίτερα προσαρμοστική και αυτό συνδυάζεται με το γεγονός ε, των οικονομικών περιορισμών ε, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Από την άλλη μεριά, η βιωσιμότητα αναφέρεται, τα ΑΕΠ ε, συνεχίζουν να βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα και υπάρχουν ακόμα τροτότητες απέναντι στις αντιδράσεις της αγοράς. Καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι για το 2018 ε, ενδείχνεται ουδέτερος δημοσιονομικός προσανατολισμός, ε, αλλά ε, συνδυασμένος με περισσότερες επενδύσεις. Η συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες είναι επίση ε, κάτι που μας απασχολεί και η ανοιξιάτικη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, φαίνεται να δείχνει ότι υπάρχει επιδείνωση στον τομέα αυτών. Από την άλλη μεριά, οι απαιτήσει ε, του Συμφώνου Σταθερότητας και ανάπτυξη φαίνεται να δείχνει ότι θα πρέπει να έχουμε πιο αυστηρούς κανόνες. Βρισκόμαστε όπως και να έχει κοντά σε ουδέτερο δημοσιονομικό προσανατολισμό και αυτό δεν είναι κάτι που αμφισβητούμε. Ιδανικό όμως ε, θα θεωρούσαμε εμείς ε, να ακολουθήσουμε ε, τους ρόμβους που βλέπετε εδώ πέρα, τους μη κόκκινους ρόμβους. Οι χώρες που έχουν ξεπεράσει ε, τους μεσοπρόθεσμους στόχους τους, εκμεταλλεύονται τις δημοσιονομικές δυνατότητες και ε, έχουν ανάπτυξη περισσότερη από την αναμενόμενη. Και η θέση αυτή σχετίζεται ακριβώς με τους μεσοπρόθεσμους στόχους τους. Εντύπωση εδώ προκαλεί ότι η κατάσταση είναι παρόμοια σε αρκετές χώρες ε, και η ρυθμή ανάπτυξης, αλλά το επίπεδο βιωσιμότητας και της ύφεσης ε, στην οικονομία διαφέρει. Ο ρυθμός ε, όμως που η παραγωγή ξεπερνάει τις ε, δυνατότητες, το δυναμικό, ε, είναι περίπου ο ίδιος, το ίδιο ποσοστό. Εξετάζουμε λοιπόν όσον αφορά τους μεσοπρόθεσμους στόχους τι συνέπειες έχει αυτό για κάθε χώρα. οι εθνικές πολιτικές ε, δεν ε, οδηγούν απαραίτητα στο βέλτιστο αποτέλεσμα για την Ευρωζώνη στο σύνολό τη και αυτό νομίζω ότι αναγνωρίστηκε όταν ε, συντάχθηκε η συνθήκη του Μάστριχτ. Αναγνωρίστηκε όμως ότι εφόσον οι χώρες διέφεραν τόσο πολύ μεταξύ τους έπρεπε να έχουν και διαφορετικές δημοσιονομικέ πολιτικέ. Επίση, οι χώρε ήθελαν να έχουν λέγην στον τρόπο διαμόρφωση των πολιτικών του. και το ε, αποτέλεσμα spillover, δηλαδή η μετάδοση πρακτικών από μια χώρα σε μια άλλη, δεν παίζουν ε, πολύ ρόλο σε καλούς ε, οικονομικούς καιρούς, αλλά στις μέρες μας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και οι ισχυρές και οι ασθενείς οικονομίες θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι αυτό το spillover Ε, έχει σημαντικές επιπτώσεις ε, και οι δημοσιονομικοί κανόνες επικεντρώνονται στο ότι δεν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ευρωπαϊκή διάσταση, έπαιζε περισσότερο ρόλο όταν υπεγράφει ε, η συνθήκη του Μάστριχτ, κάτι που μας φέρνει πάλι στο παρόν δίλημα. ότι κάποιες χώρες δεν θεωρούν οι ίδιες ότι χρειάζονται δημοσιονομική μεγέθυνση ενώ οι κανόνες ε, του συμφώνου απαιτούν ε, περισσότερη ε, σταθεροποίηση. Δύο τρόποι υπάρχουν μόνο να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Καταρχάς να το αναγνωρίσουμε και να έχουμε περισσότερο εθελοντικό συντονισμό μεταξύ των χωρών που έχουν ξεπεράσει τους μεσοπρόθεσμους στόχους τους αλλά και να έχουμε περισσότερη δημοσιονομική ολοκλήρωση, όπως συζητήθηκε και όπως προτείνεται στην ε, ε, έκθεση των πέντε προέδρων ε, του 2015. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ο πρόεδρος, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Και τώρα να αρχίσουμε την συζήτηση με τους βουλευτές. Ο κύριος Μπάλτσενε ο πρώτος συνάδελφος. Ο κύριος Πουρχαρτ Πάλ, σε ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για αυτήν την ενδιαφέρουσα πρώτη έκθεση σχετικά με τον ε, δημοσιονομικό προσανατολισμό της Ευρωζώνης. Εμείς από το ΕΛΚ ε, γενικά είμαστε αρκετά επικριτικοί όσον αφορά ε, τον συνολικό υπολογισμό. Η όπως ε, λέει ο συνάδελφος ο Γκούναρ Χεκμαρκ. Αν ε, βάλει κανείς τα πόδια στο ψυγείο ε, και το κεφάλι στο φούρνο, μπορεί πάλι η μέση θερμοκρασία να είναι η σωστή. Και παραπέμπουμε στην υποχρέωση να τηρούνται οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δεν Μπορούμε όμως να ξεφύγουμε από το γεγονός ότι τελικά κάθε κράτος μέλος ε, είναι υποχρεωμένο να κάνει τη δουλειά του και να τηρεί τους κανόνες. Είμαστε ευγνώμονες ε, και για αυτό που είπατε ε, και περιμένουμε να δούμε τις εργασίες σχετικά με το δεύτερο τμήμα της εντολής του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου να εξετάζει την τήρηση των κανόνων στα κράτη-μέλη. Είπατε ότι για το 2017 και 2018 θα έχουμε μια ελαφρά δημοσιονομική μεγέθυνση, ενώ εσείς από το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θεωρείτε ότι ουδέτερος ε, δημοσιονομικός προσανατολισμός ενδείκνυται. Εγώ πρόσεξα στην ανάλυση σας ε, ότι βλέπουμε και μείωση των ε, χρεών, αλλά λόγω της γύρανσης ε, του πληθυσμού στην Ευρώπη θα έχουμε αυξημένη πίεση στους ε, δημόσιους προϋπολογισμούς. Και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει εξέταση της δυνατότητας αποπλήρωσης χρεών των κρατών μελών. Και αυτό είναι θέμα που συνδέεται και με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Έχω κάποιες ακόμα παρατηρήσεις. Ε, καταρχάς, σταθεροποίηση του προϋπολογισμού. Ε, έχει ασκηθεί η πίεση ώστε κάποια κράτη-μέλη να αυξήσουν τις δαπάνες τους. Πρόκειται για τις χώρες που ήδη χρωστούν πολλά χρήματα ή που ε, έχουν και την ε, μεγαλύτερη γέννηση του πληθυσμού, όπως είναι η δική μου χώρα, η Γερμανία. Πώς ε, μπορούμε να αποφύγουμε να ασκήσουμε βραχή, πρόθεσμη δημοσιονομική πολιτική και κοντόφθαλμη δημοσιονομική πολιτική. Και επίσης πώς μπορείτε να διασφαλίσετε παρά τις αυξημένες δαπάνες που προβλέπονται για την φροντίδα των ηλικιωμένων, Πώ μπορούμε να αποφύγουμε αυτό να έρθει σε σύγκρουση με την απέτηση για υψηλότερου μισθούς. Ευχαριστώ πολύ. Dr. Balz, thank you for your remarks. They are very well taken. If I may begin with the the final points, obviously the concerns about the longer-term future are very relevant in this context.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 Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Δεν ξέρω ότι είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, έχουμε ίσως φτάσει δίπλα σε ένα κονσένσους ε, σε σχέση με αυτά που λέει η Κομισιό, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όλα αυτά τα όργανα αναγνωρίζουν ε, ότι κάποια πρόοδος έχει επιτελεστεί. Δεν είμαστε στο 2014 ή 2015 τώρα. Έχει γίνει κάποια πρόοδος και όσον αφορά την ανάπτυξη, την οικονομική μεγέθυνση κυρίως και μερικές χώρες τουλάχιστον έχουν μπει σε μια νέα φάση με τα προγράμματά τους. Η Ισπανία έχει γίνει μια ιστορία επιτυχίας. Υπάρχουν πάρα πολλά χαρακτηριστικά που υπονοούν ότι υπάρχουν τρόποι να υπερνικήσουμε την απεσιοδοξία που είχαμε, που εν μέρει οφειλόταν σε την υποτίμηση ε, των, της, του αρνητικού αντικτύπου που είχε η εξυγίανση το 2011 ως 2013 πάνω στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Αν δούμε αυτή τη φάση θα δούμε επίσης ότι ε, η, η, η διοίκηση είχε υποτιμήσει τον αντίκτυπο του spillover Βεβαίως ε, δεν πρέπει μόνο σε αυτό να μένουμε, αλλά νομίζω ότι βασικό επιχείρημα για προσαρμογή των δημοσιονομικών πολιτικών είναι το γεγονός ότι οι πολιτικές δεν μπορούν να κάνουν περισσότερα. Είχαμε μια νομισματική πολιτική βολική και ο χρόνος αυτός ε, χρησιμοποιήθηκε για να προετοιμαστεί κάποια ανάκαμψη αλλά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε πάνω σε αυτές τις πολιτικές. Θα έχουμε ε, το θέμα των επιτοκίων που θα μας απασχολήσει στο μέλλον και θα πρέπει να σκεφτούμε τις επενδύσεις σε ευρωπαϊκές χώρες ε, με το παρόν επιτόκιο, χωρίς ε, ε, τον αντίκτυπο, τον αρνητικό του spillover πάνω στην νομισματική πολιτική. Νομίζω το μείγμα πολιτικής είναι σημαντικό και έχουμε τη συνθήκη του Μάστριχτ. Βεβαίως, βάσει των εθνικών κανόνων δεν μπορούμε μόνο να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά τα εθνικά κοινοβούλια θεωρούν ε, την πολιτική, τη δημοσιονομική ως αρμοδιότητα εθνική και είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να υποστηρίξει κανείς ότι αυτό, ε, η πτική αυτή μπορεί να στηρίξει ένα πιο σταθερό ευρώ και υπάρχουν επιπτώσεις στην παρούσα φάση. Αυτό μπορώ να πω για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τρεμόζα. Καλώς ορίσατε αγαπητέ καθηγητά στην Οικονομική Κοινοβουλευτική Επιτροπή μας. Ενδιαφέρον το κείμενό σας. Έχω κάποιες ε, ερωτήσεις. Θυμάμαι τύπου το 2009 ο Ζουμπίνη ότι το χρέος θα είναι η μητέρα όλων των φουσκών και λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση σας όσον αφορά τη βιωσιμότητα του κρατικού χρέους στην Ευρωζώνη και γενικά για όλες τις χώρες Αναρωτιέμαι, μήπως το τέλος του προγράμματος του QE που θα έρθει σε δύο χρόνια, μήπως θα έχει ή δεν θα έχει επιπτώσεις σημαντικές μακροπρόθεσμα σε αυτή την ανάλυση και βιωσιμότητα του χρέους. Γιατί αν ξαναγυρίσουμε στο προηγούμενο σενάριο του 2010 και 2011 Οπότε είχαμε σημαντικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την εξυπηρέτηση του χρέους. Τι λέτε, τι προγνωστικά κάνετε. Θα πρέπει να περιμένουμε πολύ σημαντικές επιπτώσεις, μια που η ποσοτική χαλάρωση δύο χρόνια τερματίζεται. Άλλη μου ερώτηση, δεύτερη. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε την κατάρτιση του εθνικού προπολογισμού όσον αφορά τι δαπάνε, τόσο ώστε οι κυβερνήσει να επενδύουν. Για πετε μα τη γνώμη σα σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειαζόμαστε εναρμόνιση, την ανάλυση κόστους οφέλους των κρατικών επενδύσεων, γιατί το Κοινοβούλιο πάντοτε λέει ότι θα πρέπει αυτό να γίνει. Επιμένουμε, επιμένουμε προς τα κρατημέλη θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις για τα αεροδρόμια. Και οι χώρες, από την άλλη μεριά, επενδύουν πάρα πολλά χρήματα σε πάρα πολύ γρήγορα τρένα που κυκλοφορούν όμως άδεια ή σε αυτοκινητοδρόμους που καταλήγουν επίσης άδεια. Μήπως πρέπει να κάνουμε κάποια εναρμόνιση των μελετών κόστος κόστος-οφέλους στην Ευρώπη και έτσι να λάβουμε υπόψη τις άρεστες πρακτικές για τις κρατικές επενδύσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much for your remarks, uh, Mr. Um, Ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ τον συνάδελφο Λουβίνη και έχει δίκιο ότι το δημόσιο χρέος αποτελεί αιτία πολλών προβλημάτων ε, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη βλέπουμε ότι ε, έχει αποδειχθεί πολύ δύσκολο να ε, μειωθεί το δημόσιο χρέος, ενώ είδαμε ότι σε χώρες με υψηλό ιδιωτικό χρέος ήταν πιο εύκολο, όπως είδαμε στην Ιρλανδία και στην Ισπανία. Ήταν πιο εύκολο να λυθούν τα προβλήματα όταν πρόκειται για ιδιωτικό χρέο. Το δημόσιο χρέο είναι σημαντικό πρόβλημα και δεν θα έλεγα ότι προβλέπουμε δυσκολίες, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Είδαμε τι έγινε το 2012 στην Ιταλία και την Ισπανία. Νομίζω όμως ότι προχωρήσαμε όσο μπορούσαμε για να σταθεροποιήσουμε την συνεκτικότητα των ε, επιτοκίων ε, στα δημόσια ομόλογα. Θα πρέπει να θυμόμαστε άλλωστε ότι χρησιμοποιείται συγκεκριμένη κλίδα για την ε, αγορά ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βλέπουμε όμως να υπάρχουν τροτότητες από καιρό σε καιρό και είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε ένα σύστημα και αυτό με φέρνει στη δεύτερη σας παρατήρηση σχετικά με τις επενδύσεις. Φυσικά υπάρχουν πρότυπα για τις επενδύσεις και αυτό που είδαμε στο σχέδιο Juncker είναι ότι με περιορισμένη ποσότητα κρατικών εγγυήσεων θα μπορούσαμε να πετύχουμε μόχλευση και να δημιουργήσουμε ζήτηση για ε, επενδύσεις υψηλής ποιότητας ε, στην Ευρώπη. Τα κριτήρια λοιπόν για την απόδοση όσον αφορά την αναλογία κόστους όφελους ε, είναι πιο κρίσιμη από ό,τι ήταν στο παρελθόν. αλλά σίγουρα γίνεται πολύ καλή δουλειά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και νομίζω ότι προχωράμε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μαρίζα Ματίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την έκθεσή σας. Υποστηρίζετε ότι η δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωζώνη είναι προνόμιο των εθνικών κυβερνήσεων. Και νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε εδώ στο Κοινοβούλιο ότι αυτό δεν είναι τόσο απλό το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διακυβέρνησης δημιουργήθηκε και ορίζει τις προϋποθέσεις για τη δημοσιονομική πολιτική των κρατών μελών πέρα από τα όρια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ε, και η ε, επέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και άλλων θεσμικών οργάνων ε, δεν περιορίζεται στη δημοσιονομική πολιτική. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δημοσίων πολιτικών όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, η φορολογική πολιτική και η αγορά εργασίας. Όπως και να έχει, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποιες από τις ιδέες που αναφέρατε και που συμπεριλαμβάνονται στην εκθεσή σας. Γενικά λέτε ότι Μπορούμε έτσι να οδηγηθούμε σε μια υγιή συγκέντρωση του ε, χρέους ε, και έτσι σε καλύτερο δημοσιονομικό προσανατολισμό. Δεν μπορώ όμως να καταλάβω ποια είναι η ανεπαρκής χρήση δημοσιονομικής πολιτικής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμένα μου φαίνεται προφανές ότι οι πολιτικές λιτότητες υπονόμευσαν πολύ σημαντικά την δημοσιονομική πολιτική. Μόλις αναφέρατε την περίπτωση της Πορτογαλίας, ε, και εγώ Πορτογαλίδα είμαι, και δεν ε, αναφερθήκατε στις επιπτώσεις του προγράμματος ε, της Τρόικας. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ευρωζώνη παλεύει με το θέμα αυτό για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα και δύο παράγοντες έχουν συμβάλει στην τρελή αυτή κατάσταση. Καταρχάς, ε, η ε, ρύθμιση της αγοράς εργασίας ε, και οι δημοσιονομικές πολιτικές. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η θέση σας για τα δύο αυτά θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Μαρίσα Ματίας, για τις παρατηρήσεις σας, παρόλο που ε, είχαν κριτική. Νομίζω θα πρέπει να διακρίνουμε σαφώς ανάμεσα στην κατάσταση όπου χώρες και προγράμματα όπου ο βαθμός παρέμβασης είναι πιο λεπτομερής ε, στην, ε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα ήθελα να σας πω ότι στον δικό μας το Συμβούλιο το Δημοσιονομικό δεν ε, εξετάζουμε τις χώρες, ε, τα προγράμματά τους, ε, διότι η εποπτεία είναι πάρα πολύ λεπτομερής και δεν είμαστε εμεί για να αυξήσουμε την εποπτεία και για παρέμβαση. Είναι μια διαφορετική κατηγορία. Όταν υπάρχουν ζημίες και έχετε πρόσβαση στις αγορές, τις χρηματοοικονομικές, είναι κατανοητή κατάσταση και, από, και βάσει της πείρα στη δική σας χώρα είναι δυνατόν να βγείτε από ένα τέτοιο πρόγραμμα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα βεβαίως με μεγάλες θυσίες το κάνατε το κάνατε ενώ είχατε ε, διαφορετικές ε, κυβερνήσεις στη χώρα σας. Δεν το θεωρώ αυτό ως αποτυχία. Βεβαίως υπάρχει ένα όριο ε, χρονικό για τις παρεμβάσεις αυτές για να θέλει κανείς να διατηρήσει εθνική κυριαρχία. Να εξετάσετε την εμπειρία πολλών άλλων χωρών έχουν μια φιλελεύθερη ε, στάση, ε, ίσως πάρα πολύ φιλελεύθερη αν ε, δείτε πώς εφαρμόζουν τα στάσεις τις σχετικές ειδικά με κάποια χώρα. Ε, και βλέπετε ότι μειώνεται η συμμόρφωση και είναι βεβαίως ορισμένες εθνικές θέσεις αυτές. Εγώ προσωπικά λυπούμαι γι' αυτό, αλλά δεν μπορεί κανείς να αφισβητήσει ότι η δημοσιονομική πολιτική είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό μια εθνική αρμοδιότητα και δεν μπορούμε να πείσουμε τις χώρες αυτές ε, για την σημασία των ε, επιπτώσεων spillover των πολιτικών τους. Βεβαίως και εγώ ε, κατέκρινα στο Συμβούλιο ε, για την 2011 με 2013 τα προγράμματα εξυγίανσης ίσως ήταν υπερβολικά, ε, ίσως προχωρήσαμε πολύ μακριά, πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Βεβαίως συζητούμε αυτό τον προσανατολισμό, το, την επίπτωση, το fiscal stance για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Σβέν Γίγκολτ είναι εδώ. Ο κ. Σκόμπερν. Πάρα πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ μαζί μας. Πολύ ενδιαφέροντα όσο μας είπατε. Ήσασταν σε εκείνη την ανοιχτή συνάντηση των συνονισμών της 14ου, 12ου του 16 και τον Ιούνιο του 2017 συζητηθεί η έκθεσή σου χρόνο το fiscal stance για την Ευρωζώνη και είχατε πει ότι το 2018 θα έχουμε ένα fiscal stance ουδέτερο, το οποίο θα είναι το πιο δόκιμο για το σύνολο της Ευρωζώνης. Και τέτοιο fiscal stance θα αφορά τις ε, εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να έχει μια κοινή φορολογική πολιτική για όλα τα κρατημέλη. Όμως, αυτά τα οποία είπατε, με τα οποία και συμφωνώ, αποκλίνουν τις απόψεις της Επιτροπής και τις επιθυμίες της. Είχαμε δε διαβάσει στον τύπο την περσμένη εβδομάδα όσον αφορά την τέταρτη οδηγία κατά του ξεπλήματο χρήματο, ότι θέλουν να σταματήσουν την φοροδιαφυγή με αυτά τα μέτρα. Όμως, σύμφωνα με τη δική μα νομολογία, είναι υποχρεωτικό να έχουν φορολογικές απαλλαγές συμμετοχή γιατί η φοροδιαφυγή είναι παρανομή αλλά η φορολογική ελάφρυνση μέσω τέτοιων μέτρων δεν είναι κάτι το παράνομο. Τα είχα πει αυτά στην Επίτροπη εβδομάδα. Και συμφωνήσαμε ότι, ότι θα πρέπει να κατασταλεί η φοροδιαφυγή. Αλλά δεν νομίζω ότι κατάλαβε τη διαφορά φοροδιαφυγής και φορολογικών ε, μέτρων αποφυγής παραβολιβαριάς φορολογίας. Ε, ε, δηλαδή θέλει η Κομισιόν να μαζέψει χρήματα από όσο γίνεται. Ε, εντάξει, ο Άνταμ Σμιθ Σκοτσέζος ήταν, ε, αλλά φαντάζομαι και εσεί συμφωνείτε με αυτό που λέγει. Έχουμε μπερδέψει τώρα το θέμα δημοσιονομικό με το φορολογικό λόγω του, ε, των, των όρων. Άλλο πάει να πει στα Ιταλικά και άλλο στα Αγγλικά, τέλος πάντων. Αλλά ας απαντήσει ο φιλοξενούμενος μας. Σας ευχαριστώ κύριε Κόμμα. Αυτό ήθελα να πω και εγώ και με προλαβεί ο πρόεδρος. Υπάρχει αυτή η διάκριση για αυτό το θέμα της ε, φορολογικής ε, εναρμόνισης. Είναι θέμα μακροοικονομικό περισσότερο, ξέρετε. Θα πρέπει και αυτό να μας απασχολήσει. Αλλά και βέβαια η φοροαποφυγή είναι ένα σημαντικό θέμα. Τώρα η σχέση με τις μακροοικονομικές πολιτικές ε, είναι τέτοια που θα μπορούσαμε να κάνουμε εναρμόνιση και να έχουμε πιο αποτελεσματική νομοθεσία γιατί ακριβώς υπάρχουν θέματα πολύ διφορούμενα όσον αφορά στο τι γίνεται όσον αφορά τη φορολογία των εταιριών και για την φοροδιαφυγή να εγκυμονούνται κίνδυνοι εάν αυτά τα μπερδεύουμε. Fiscal stance δεν σημαίνει ότι θα πρέπει οι πολιτικές να είναι ίδιες. Μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε χώρα, στη δυοσημότητα του χρέους, την οικονομική συγκυρία, τη σταθεροποίηση της κάθε οικονομίας. Να ποια είναι η σχέση, η ανυπαρξία σχέσης μεταξύ των δύο. Και εκεί που δεν πήγαμε καλά στο παρελθόν, ήταν το ότι οι κοινέ πρωτοβουλίες παρά ήταν κοινέ, παρά ήταν ίδιες για περισσότερες χώρες. 2007-2008 για τη χρηματοπιστωτική κρίση, οι περισσότερες χώρες είχαν επεκτατική πολιτική και το συνέχισαν. Οπότε τελικά η οικονομία τους αδυνάτησε. Άρα το παράκαναν με τις σχετικές συστάσεις. Μετά είπε η Κομισιόν, έχουμε τώρα την ανάκαψη και πάμε στο 0,5% για όλους. Οπότε έτσι εκτίθενται οι πιο αδύναμες δημισιονομικά χώρες. Και μετά στην περίοδο της οικονομικής συρρήκνωσης στριμώχνονται πολύ. Δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο για όλους. Επιβάλλεται η διαφοροποίηση. Και φυσικά θα πρέπει να είναι δίκαιοι οι κανόνες για την εναρμόνιση, αλλά και για την ε, αντιμετώπιση της φοροαποφυγής. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Ε, στην πρώτη έκθεση του οργάνου σας, για πρώτη έκθεση απογοητεύομαι. Ε, το Συμβούλιο είναι ανεξάρτητο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αυτό δεν το βρίσκουμε στην έκθεσή σας και δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη πρόταση. Κι όμως ε, η Γερμανία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια για να χρηματοδοτεί δημόσιες επενδύσεις ε, στις εθνικές υποδομές, πράγμα που θα, θα έκανε πιο δυναμική την Ευρωζώνη. Επίσης, ε, τις ελλείψεις της Ευρωζώνης δεν τις κατακρίνεται τις σταθερές ιστοτιμίες που αποτρέπουν, που παρεμποδίζουν την προσαρμογή των ισοτιμιών μεταξύ των χωρών. Τίποτα για την υπερχρέωση των κρατών μελών που ίσως είναι, θα επιβαρύνει τις μελλοντικές γενναίες. Για το πρόβλημα της δημοσιονομικής υπερχρέωσης, μήπως σκοπεύετε στην επόμενη έκθεση να προτείνετε συγκεκριμένες προτάσεις ε, για να μπορέσετε να ελευθερώσετε τις χώρες από αυτήν την δουλεία ε, σε παγκόσμιες αγορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μονού. Νομίζω ότι είμαστε ανεξάρτητοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως δεν το βλέπετε, δεν το διαπιστώνετε στην έκθεση. Βεβαίως, ε, συμφωνούμε με την Κομισιόν για το 2018 και η ανάλυση ε, δείχνει ότι υποστηρίζουμε αυτή τη σύσταση. Βεβαίως, ε, ε, συμφωνούμε με την Κομισιόν για την ώρα, δεν την κατακρίνουμε. Ε, για στη φάση αυτή συμφωνούμε με την Κομισιόν. Αλλά δεν ε, ασκεί καμία πίεση η Κομισιόν πάνω μας και η γραμματεία μας είναι ανεξάρτητη και δεν παίρνει οδηγίες από την Κομισιόν. Ε, καμία πίεση δεν ασκείται πάνω μας από ε, την Κομισιόν, πάνω στους συναδέλφους ε, που είναι καθηγητές, πανεπιστημιακοί και έχουν την δική, δική τους άποψη. Νομίζω ότι στην επόμενη έκθεση θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες για τις μεμονωμένες χώρες και τότε Ίσως θα δούμε ποια είναι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις χώρες και στην Κομισιόν και πώς το σύστημα έχει γίνει τόσο δύσκολο και είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε και τότε εκεί θα υπάρχει κάποιο πεδίο ε, για κάποια συγκεκριμένη πρόταση και ίσως και για κάποια κριτική, αλλά ακόμα δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Βεβαίως εσείς ε, κατακρίνατε την ε, κατάσταση. Υπάρχουν ε, βεβαίως άλλα προβλήματα σε ορισμένες χώρες. Δεν νομίζω ότι μπορούν να επιληθούν τα προβλήματα αυτά με την, Ευρωπαϊκή, με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Βεβαίως υπάρχει ε, μια διαδικασία η οποία εξετάζει τις ανισορροπίες, η οποία υφέρπει για την ώρα, δεν χρησιμοποιείται, είναι σε λανθάνουσα κατάσταση. Ε, παρακολουθούμε τους δείκτες, τους παρακολουθεί και η Κομισιόν, αλλά η κατάσταση είναι πολύ πιο ε, δύσκολη από, από ό,τι φαίνεται με το Σύμφωνο Σταθερότητας. Νομίζω ότι όταν βλέπουμε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες είναι νομίζω ένα τομέα, ένα σκέλος το οποίο έχει παραβλέφθηκε μέσα στο σύνολο των ανισορροπιών της οικονομίας. Βεβαίως θα συνεχίσουμε ε, και θα βασιζόμαστε στους μηχανισμούς οι οποίοι υπάρχουν και θα τους χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ε, βεβαίως υπάρχουν ε, ε, ορισμένες χώρες οι οποίες έχουν αρκετή εξωστρέφεια και έχουν παρουσιάσει καλά αποτελέσματα με τις εξαγωγές τους. Η Γαλλία έχει νομίζω ένα πλεόνασμα ως προς το τρέχον ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις στις τελευταίες στιγμές, ένα λεπτό μας μένει μόνο όμως. Αλλιώς μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και επικοδομητική. Εγώ προσωπικά βρήκα πολύ πιστική και την εκτίμηση της κατάστασης της ανάκαμψής μας. Βλέπουμε μια κυκλική ανάκαμψη με μια σειρά στοιχείων που δείχνουν ότι απαιτείται ακόμη πολλή δουλειά. Και χρειάζεται αποτελεσματικός συντονισμός. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ε, τα εργαλεία για να έχουμε τέτοιο, τέτοια αποτελεσματική εφαρμογή και δεν ξέρω αν τα εργαλεία για τις μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες, αν μπορούν ε, αυτά να αποτελέσουν ε, εργαλεία για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Φαίνεται να είναι απαραίτητος λοιπόν ο δημοσιονομικός συντονισμός που προτείνετε εσείς, αλλά το ότι είναι απαραίτητος δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι και πολύ δύσκολος. και βλέπουμε ότι κάποια κεντρικά συστήματα της δημοσιονομικής πολιτικής και ε, κάποια εθνικά στοιχεία και η ανάγκη να συντονιστούν τα πρώτα με το δεύτερα είναι κάτι που θα πρέπει να εξετάσουμε. Το σχέδιο Juncker αποτελεί μία προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να βελτιώσουμε την ποιότητα, όχι μόνο την ποσότητα στον ε, τρέχοντα τριμερή διάλογο. Διότι το θέμα δεν είναι μόνο ε, οι δημοσιονομικές ε, στατιστικές, αλλά πρέπει να εξετάσουμε και τους επιμέρους τομείς και τι γίνεται εντός του κάθε τομέα. Είναι λοιπόν πολύπλοκο και δύσκολο το έργο μας. Αλλά νομίζω ότι πολλά υπόσχεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και ότι μπορεί να συμβάλλει σε μία σοφή προσέγγιση ε, των προβλημάτων αυτών. Έχουμε λοιπόν ε, διάφορους παράγοντες εδώ πέρα και θα χαρώ πολύ και στη συνέχεια να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο σας ε, ώστε να έχουμε δημοκρατική διαφάνεια και πιο αποτελεσματικό δημοσιονομικό συντονισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. So, uh, two of suspension. Δύο λεπτά διακοπή για να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο σημείο 6 της ημερησίας διάταξης. Έχουμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Πάνω στην νομοθετική πρόταση οδηγίας σχετικά με την ενδυνάμωση των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών προκειμένου να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τη σχετική νομοθεσία και να διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Όπως γνωρίζετε αυτό το θέμα είναι πολύ επίκαιρο διότι αποτελεί αντικείμενο συναπόφασης. Επικροτούμε λοιπόν την πρόταση αυτή επειδή ε, καλύπτει πολύ σημαντικά θέματα. Η συγητής είναι ο κύριος Σφάμπ. και γνωρίζετε ότι είχαμε οργανώσει σεμινάριο για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας ενημερώσω επίσης ότι η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου έχει ξεκινήσει τις εργασίες πάνω στο θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της Μαλτέζικης Προεδρίας και συνεχίζει τις εργασίες της ε, τώρα υπό την Εστονική Προεδρία. Κύριε, Προ... έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για πρώτη φορά αυτήν την πρόταση οδηγίας σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού ΣΥΝ. Όπως είπε ήδη ο Πρόεδρος, πρόκειται για σημαντική εξέλιξη ενός κεντρικού τομέα των ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων. Το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα υποβάλλει αυτή την πρόταση δείχνει δύο πράγματα. Καταρχάς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπιστεύεται το Κοινοβούλιο, διότι είναι δεύτερη νομοθετική πρόταση στον τομέα του ανταγωνισμού που περνά από το Κοινοβούλιο. Και μαζί με του ε, σκιώδεις εισηγητές, με του οποίου είχα ήδη συνάντηση, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε στην ε, εμπιστοσύνη αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, ε, κύριε Πρόεδρε, στον τομέα αυτών υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούν και πρέπει να βελτιωθούν. Πρόκειται για τομέα ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων όπου μάλλον υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατότητα επέμβασης από πλευράς ε, της Ευρώπης. Από την άλλη, ε, χρειαζόμαστε και ένα πάρα πολύ ευέλικτο μέσο. Και έτσι έχουμε το δίλημα ότι από τη μία θέλουμε ασφάλεια δικαίου για τους ε, εμπλεκόμενους και από την άλλη θέλουμε ευελιξία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το πώς θα το πετύχουμε αυτό σίγουρα θα αποτελέσει το επίκεντρο των συζητήσεων μέσα στους επόμενους μήνες. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι δεν επηρεάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το θέμα αυτό. Ε, το θέμα είναι απλά η εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 από πλευράς των κρατών μελών. Από την άλλη θα υπάρξουν σίγουρα και τομείς επικάλυψης όπου οι αρχές ανταγωνισμού των ε, κρατών μελών θα πρέπει να εφαρμόσουν ευρωπαϊκό δίκαιο και γι' αυτό θα πρέπει αυτό να γίνει επιτυχώς. Από τη μία θέλουμε ενότητα όσον αφορά το δίκαιο, από την άλλη θέλουμε οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού να έχουν επαρκές περιθώριο ώστε να μπορέσουν ε, να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους με ομαλό τρόπο. Η αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού από τις, ευρωπαϊκές, ε, από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού είναι κάτι που θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα ωφελήσει και τις επιχειρήσεις. Έτσι θα εξαλειφθούν τα εμπόδια στην εσωτερική αγορά και θα διασφαλιστεί περισσότερη ασφάλεια δικαίου για τι επιχειρήσει. Γενικά νομίζω ότι μπορούμε να επικροτήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει το Κοινοβούλιο να εξετάσει αναλυτικά ως νομοθέτης. Το πρώτο θέμα που είναι σημαντικό για μένα είναι το άρθρο 3.3 πρότασης. Αναφέρεται ότι υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, είναι πολύ σωστά όλα αυτά, ε, αλλά ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων ήδη υπάρχει και γι' αυτό είναι αρκετά προφανές ε, αυτό που λέει το άρθρο 3. γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρετε πιο συγκεκριμένα τι σημαίνει ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων στο δίκαιο ανταγωνισμού. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να, να, να βρούμε τουλάχιστον κάποιες ε, ε ορθές πρακτικές ε, που να είναι σχετικές με το θέμα αυτό. Το ίδιο θέμα ισχύει και για το αν όλα αυτά θα πρέπει να ισχύουν και για ασφαλιστικά μέτρα και σε άλλες διαδικασίες. Πάντως ε, είναι θέματα που θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Δεύτερη παρατήρηση αφορά το άρθρο 8 ε, και τα αιτήματα παροχής ε, πληροφοριών. Πιστεύω ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να αρνηθούν να παράσουν πληροφορίες, ώστε να μην αυτοενεχοποιούνται και θέλουμε από τη μία αποτελεσματική εφαρμογή του ε, δικαίου περί ανταγωνισμού και από την άλλη θέλουμε και σεβασμό των αρχών ε, του κράτους δικαίου. Θα πρέπει λοιπόν εδώ επίσης να βρούμε τη σωστή ισορροπία εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, αναφέρθηκα ήδη στα ασφαλιστικά μέτρα, στα προσωρινά μέτρα. Ενδιαφέρον είναι ότι όσον αφορά την ψηφιακή αγορά έχει ξεκινήσει συζήτηση μήπως θα πρέπει να είναι ε, πιο συχνά δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινά μέτρα. Τα μέτρα αυτά προβλέπονται για τις αρχές ε, των ε, κρατών μελών. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει νόημα να μην υπάρχει καμία δυνατότητα για τις ευρωπαϊκές αρχές ε, να παρέμβουν. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε πώς το ευρωπαϊκό επίπεδο θα συντονιστεί με το εθνικό. Τρίτον, οι διαδικαστικές απαιτήσεις που ρυθμίζονται εδώ μήπως θα πρέπει να διαβρινθούν και να έχουμε εδώ δεσμεύσεις έχουμε τις συμφωνίες μεταξύ των καρτέλ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι διαδικασίες αυτές ε, διέπονται από αυτά τα ελάχιστα πρότυπα. Τέλος, έχουμε το θέμα των ε, χρηματικών προστήμων. Ε, υπάρχει το ανώτατο όριο του 10% και εφόσον στην πράξη ισχύει αυτό, γιατί να μην έχουμε ένα ενιαίο όριο για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό νομίζω θα αποτελούσε σημαντική απλούστευση στο θέμα αυτό, την οποία θα πρέπει τουλάχιστον να εξετάσουμε. Επίσης, όσον αφορά την, ε, την κοινή γεωργική πολιτική, πώς θα πρέπει να εξετάζουμε τις επιμέρους χώρες ή πώς πρέπει να ετοιμάσουμε τα γενικά ε, επίπεδα και θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι ε, οι παραβαίνοντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πριν την επιβολή προστίμου να αποκαταστήσουν την κατάσταση. Ε, κάτι που ε, θα αποζημιώσει πιο γρήγορα τον καταναλωτή. Όσον αφορά τις γενικές ε, αρχές, ε, νομίζω ότι είναι ισορροπημένη η πρόταση οδηγίας. Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε όταν ένας βασικός μάρτυρας υποβάλλει έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι αρμόδια, πώς μπορεί αυτό με ασφαλή τρόπο να μεταφερθεί στις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού, να έχουμε δηλαδή μια ενιαία θηρίδα, ένα one-stop shop. Πάντως, γενικά νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα λύνονται ε, με πολύ ικανοποιητικό τρόπο στο πλαίσιο της πρότασης. Ε, γι' αυτό θα ήθελα απλά να αναφέρω, κύριε Πρόεδρε, ότι ε, η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί 9-10 Οκτωβρίου, τροπολογίες μέχρι τις 20 Οκτωβρίου και στις 4 Δεκεμβρίου θέλουμε να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή. και έτσι υπό την Εστονική Προεδρία πιθανότατα να καταλήξουμε σε ε, αποτέλεσμα ε, που θα, κάτι που θα ταιριάζει και με τη γραμμάτα που ε, φοράμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μας δώσατε και το χρονοδιάγραμμα. Ρεαλιστικό. Πρώτα, ο Σκιώδης σύγητης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτήν την πλήρη παρουσίαση ε, του θέματος, ε, τον συγχαίρω, διότι ε, επίσης συμπεριέλαβε όλα τα σημαντικά στοιχεία. Όλοι εδώ έχουμε διευκρινίσει με μεγάλη πλειοψηφία ότι ε, το, σχέδιο σχετικά με τον ανταγωνισμό που εγώ είχα συντάξει ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού ε, προς όφελος του ε, ανταγωνισμού και της συντονισμού. Εξ ονόματος της ομάδας μου θα θέλαμε να δούμε το πρώτο σχέδιο της έκθεσης. Εγώ χαίρομαι που ο ε, Πίτροπος ήταν ανοιχτός σε αυτό το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για την, ε, τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, για την ενδυνάμωσή τους και ελπίζω ότι τα δύο όργανα θα συνεργαστούν στενά για το θέμα αυτό. Ωστόσο τώρα θα ήθελα να τονίσω τρία θέματα για να προτείνω στον εισηγητή να τα περιλάβει στο πρώτο σχέδιο έκθεσης. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό για μας, για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ηγεσία. Θα πρέπει ε, η ανεξαρτησία της ηγεσίας των εθνικών αρχών ανταγωνισμού να υπάρχει παντού σε όλα, σε όλα τα κράτη-μέλα. το χάρη ο διορισμός των επικεφαλής δεν πρέπει να βασίζεται σε πολιτικά κριτήρια, αλλά μόνο σε επαγγελματικά κριτήρια και στην πολιτική πείρα και στην επαγγελματική πείρα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι θα πρέπει να συνδεθούν ε, με τα κατάλληλα οικονομικά μέσα. Οι οικονομικοί πόροι των εθνικών αρχών ανταγωνισμού δεν μπορούν να βασίζονται ε, στα πρόστιμα που επιβάλλονται, παραδείγματος χάρη. Έχουμε πρακτικές ορισμένα τα κράτη-μέλη που μπορούμε να χρησιμοποιούμε, βέλτιστες ε, πρακτικές, παραδείγματος χάρη, Επίσης θα ήθελα να προσθέσουμε στην χρηματοδότηση ότι το έργο των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού είναι να πάρε, δεν είναι μόνο ένας μηχανισμός ελέγχου, αλλά επίσης και μια παροχή υπηρεσίας. Ε, αυτό είναι μια εγγύηση ότι θα μπορούν να λειτουργούν σε ένα πραγματικό ανταγωνιστικό περιβάλλον και ότι κανείς δεν θα μπορεί να παραβιάσει τους κανόνες ανταγωνισμού χωρίς συνέπειες. Και τέλος θα ήθελα να τονίσω την αναγκαιότητα εναρμόνιση σχετικά με τους κανόνες καταπολέμησης της διαφθοράς και την προστασία των, των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Όλα αυτά βασίζονται στο, σε όλα το πλαίσιο των θεμάτων που εξέθεσε ο εισηγητής και νομίζω ότι με αυτές τις παρατηρήσεις θα μπορούμε να έχουμε μια πληρέστερη εισήγηση και πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σταρμπάτη από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Το ECR καταλαβαίνει την αναγκαιότητα των όσων έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός είναι να αποφύγουμε ε, την αναζήτηση του ευνοϊκότερου καθεστώτος ε, για τις επιχειρήσεις. Η κατεύθυνση που ακολουθεί η πρόταση οδηγίας μας φαίνεται πολύ λογική. το θέμα είναι πώς μπορούν οι, ευρωπαϊκές, οι εθνικές ε, αρχές ανταγωνισμού να βελτιώσουμε την εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού και να γίνει η προσαρμογή στις εθνικές ε, παραδόσεις ώστε να ανταποκριθούμε ε, στην αρχή της επικουρικότητας. Το ECR δίνει ιδιαίτερη σημασία στο ότι συχνά ε, είναι εις βάρος του καταναλωτή η δημιουργία καρτέλ και αυτό συχνά γίνεται από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό η ανεξαρτησία των ε, εθνικών αρχών ανταγωνισμού είναι η ιδιαίτερη σημασία για το ECR. Σύμφωνα με τον ΩΣΑ, το 86% των ε, επιχειρήσεων δεν έχουν σωστή μεταχείριση λόγω τη μη σωστή εφαρμογή των αρχών ανταγωνισμού. Το ECR θέλει λοιπόν ίση μεταχείριση όλων των συμμετεχόντων ε, στην αγορά. Το ECR στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι είναι απαραίτητο να αποφύγουμε την αναζήτηση του ευνοϊκότερου καθεστώτος από πλευράς των επιχειρήσεων, καλύτερη ε, βοήθεια από τις αρχές και πρόγραμμα για τους βασικούς μάρτυρες. Και δεν θέλουμε επιπλέον γραφειοκρατία στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Εμείς ευχαριστούμε. Για την άλλη τώρα, κύριος Γιέζικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να εξασφαλίσουμε τον θεμητό ανταγωνισμό θα πρέπει να λειτουργεί με εσωτερική αγορά εξ αυτού του λόγου. οπότε και θα πρέπει οι αρχές ανταγωνισμού να έχουν ε, τους πόρους, να έχουν τα μέσα, ούτως ώστε να εφαρμόζουν το κοινωτικό δίκαιο σε αυτό τον τομέα για την ομάδα των φιλελευθέρων θέλουμε να σταθούμε σε κάποια συγκεκριμένα σημεία βέβαια κάποια προαναφέρθηκαν πρώτα πρώτα είναι το θέμα των κυρώσεων που χρειάζεται να έχουν αποτελεσματικότητα θα πρέπει να αποτρέπονται από την παρανομία οι εταιρείε. θα πρέπει τα μέτρα να είναι εναρμόνιση θα πρέπει να έχουν αναλογικότητα και ταυτόχρονα να υπάρχει αναλογικότητα με το μέγεθος της εταιρεία τόσο ώστε να ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ. Οι πληρωμές επίσης είναι σημαντικό ζήτημα, οπότε θα πρέπει και εδώ να είναι οι διατάξεις στεγανές, επαναλλαγή πληροφοριών, μεταξύ των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και μεταξύ των επιμέρους εθνικών αρχών και αυτό είναι σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε την αμυροληψία, την ανεξαρτησία των αρχών και να δούμε κατά πόσον οι ερευνητικέ αρμοδιότητε των εθνικών αρχών μπορούν να αναβαθμιστούν. Τέλος, όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους αλλά και τους οικονομικούς πόρους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει όλες τις εθνικές αρχές, όλοι να λάβουν τις ευθύνε τους. Οπότε να έχουν επάρκεια προσωπικού που να έχει τις κατάλληλες δεξιότητες σε συνεργασία, Πρόεδρε, με τον εισηγητή και τους άλλους σχεδοσηγητές, θα προσφέρουμε ένα σχέδιο κειμένο, ταχαίως, και ελπίζουμε να είναι εύστοχο. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Παλώμα. Παλώμα περιμένω, δεν είναι εδώ. Σφέν Γκίγκολ για τους πράσινους. Μάλιστα. Καταρχάς, χαιρετισμούς από τον συνάδελφο Μισελ Ραϊμόν που ε, θα συνεργαστεί μαζί σας ε, κύριε Σφάπ και με τους ε, συναδέλφους. Κρίμα που δεν είναι εδώ η αριστερά, αλλά ο ανταγωνισμός είναι καπιταλιστική έννοια, οπότε ύποπτη. Θα ήθελα στο όνομα του Μισελ Ραϊμόν να σα ε, κάνω κάποιε βασικέ παρατηρήσει. Ε, Ω πράσινη στηρίζουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούμε ότι είναι καλή πρόταση και το είπαν και οι συνάδελφοι. Ανταποκρίνεται στις εμπειρίε που συγκεντρώσαμε κατά τη διάρκεια της κατοπολέμησης ε, τη νομιμοποίηση παράνομων εισόδων εθνικές αρχές ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να είναι ανεξάρτητες αρχές ε, που να εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η ανεξαρτησία και τα καθήκοντά τους ρυθμίζονται στην πρόταση αυτή και ως πράσινοι θα φροντίσουμε θέματα όπως είναι η σύγκρουση συμφερόντων και η σχέση ανάμεσα στο ε, δημόσιο συμφέρον και το ιδιωτικό συμφέρον ε, να ρυθμίζεται σαφώς. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού μπορεί να είναι αρμόδια για μια ε, υπόθεση να αποσύρεται από την υπόθεση. Ε, οι συνάδελφοι να περάσουν στην DG Comp ε, κατόπιν να μην επιτρέπεται να εργαστούν ε, στις ίδιες υποθέσεις να επανέρχονται στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και έτσι έχουμε αυτή την περιστρεφόμενη πόρτα, κάτι το οποίο ε, αποδυναμώνει την εμπιστοσύνη προς, τον, ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε και σε εθνικό επίπεδο. Είναι σημαντικό όλες οι ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού να μπορούν να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις. Ε, αυτό δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή. Πολύ σωστή λοιπόν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και επίσης σημαντικό για μας είναι η ευθύνη για τις κυρώσεις να την ευθύνη για τις κυρώσεις να την έχει το σύνολο της επιχείρησης. Ε, διότι σε μερικές περιπτώσεις βλέπουμε να προστατεύεται η μητρική επιχείρηση από τις θηγατρικές ε, και ε, έτσι να μην έχουμε τελικά αποτέλεσμα. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να είναι τόσο ισχυρά τα προγράμματα κατακελώντων. Και μία προσωπική παρατήρηση, επιτρέψτε μου, δεν είναι του Μισελ αυτή. Κύριε Σουάμπ, νομίζω ότι πρέπει να υπερασπιστείτε μια μεγάλη παράδοση, το Τσέντε Τσέσου. Ε, είναι κληρονόμος ε, του Όικεν και άλλων ε, και ο κύριος Σταμπάτη. Νομίζω θα ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για το θέμα αυτό. Άκουσα πόσο αναφερθήκατε στα θεμελιώδη δικαιώματα και αναφερθήκατε στο δικαίωμα των επιχειρήσεων να μην παρέχουν πληροφορίες. Ε, νομίζω όμως ότι και άτομα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Πιστεύω ότι τα άτομα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μην παρέχουν πληροφορίε. Οι επιχειρήσει όμω δεν νομίζω ότι πρέπει να το έχουν. Πρέπει να λογοδοτούν για την ε, για τις κακές τους πρακτικές. Νομίζω ότι οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου θα πρέπει να βρουν τη σωστή ισορροπία ανάμεσα ε, στις ε, αρχές του κράτους δικαίου και στην προσπάθεια να καταπολεμήσουμε τα καρτέλ και τις καταχρήσεις στην αγορά. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Με κανέναν τρόπο δεν θα πρέπει να ενεργήσουμε μονομερός και να θεωρούμε ότι εδώ μιλάμε για παραβίαση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου τον ε, ε, καταναλωτή που έχει υποστεί κάποια ζημιά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω πουθενά την Μπαρακάπελ ή κανέναν άλλον από τους Κιώδης. Ο Κρίστε Κέινς, ε, Διευθυντής ε, της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, είναι παρόν. Ε, σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ. Σας δίνω το λόγο, παρακαλώ. Thank you very much, President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, and for your... Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους κοιότητες εισηγητές. Πολύ ενδιαφέροντα. Όλα αυτά που λέτε. Είναι πολύ σημαντικό που εμπλέκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Επίσης το ότι έχετε εσείς κυρίες Ζερμοδιότητα είναι πολύ σωστό. Όπως ξέρετε, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικοί συνομιλητές οι εθνικές αρχές τη τελευταία δεκαετία. Όμως συμφωνούμε ότι μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα εάν έχουν τους πόρους που τους χρειάζονται. Ε, για αυτό και κάναμε και την πρόταση αυτή με τους τέσσερις άξονες την επίοικια, την εργαλειοθήκη, τους πόρους και... οπότε είπαμε ότι είναι πρόταση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έτσι να βελτιωθεί η εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού να έχουν τις ελεύθερες εγγυήσεις ότι μπορούν να έχουν ανεξάρτητες αποφάσεις οι αρχές και να μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις. Εμείς προτιθέμεθα να ακούσουμε προσεκτικά τι έχετε να πείτε με επιφύλαξη κάθε μελλοντικής αλλαγής τοποθέτησής μας. Ε, βέβαια, πάρα πολύ βασικό είναι αυτό που αναφέρθηκε για την ανεξαρτησία. Υπάρχει ευρεία συνένεση ότι αυτό είναι προϋπόθεση για ε, αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου. Ο κανονισμός ένα δεν προέβλεπε στεγανά μέτρα. Θα πρέπει να υπάρχουν τέτοια. Να μην υπάρχει α, κίνδυνος επηρεασμού των αγών αυτών από ιδιώτες ε, ή δημόσιους φορείς και παράγοντες. Στο παρελθόν διαπιστώσαμε ότι κάποιες εθνικές αρχές όποτε απειλήθηκε η ανεξαρτησία τους στράφηκαν σε εμά για βοήθεια αλλά δεν υπήρχε νομική βάση για να τους βοηθήσουμε. Οπότε θεωρούμε ότι τώρα έχουμε μια σώροπη ε, πρόταση, υπάρχουν ε, ελάχιστες εγγύησεις, δεν είμαστε υπερβολικά αυστηροί. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε τέλος πάντων για να βελτιθεί η κατάσταση τώρα όσον αφορά το δικαίωμα υπεράσπισης που θα πρέπει να είναι σεβαστά για τις εταιρείε, αλλά θα πρέπει να είναι για το μήνυμα ξεκάθαρα. Και εδώ προσπαθούμε να βρούμε ισορροπή λύση. Από τη μία μεριά έχουμε την αποτελεσματικότητα των αρχών και από την άλλη μεριά θα πρέπει να υπάρχουν εγγύησει για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Δεν θα πρέπει αυτή η ισορροπία να ανατραπεί. Και αν κάποιος προσπαθήσει με μεγάλη λεπτομέρεια να νομοθετήσει, τότε θα έρθουμε σε σύγκρουση με τις νομικές παραδόσεις των κρατών μελών. και θα διαταραχθούν οι έρευνες των εθνικών αρχοπών, το θέλουμε αυτό. Λάβουμε υπόψη και τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων που μας διευκολύνει όταν θέλουμε να παρέμβουμε για κάποιο είδου κατάχρηση εξουσίας. Οι εταιρείε θα πρέπει να έχουν κίνητρα να ζητήσουν επίκαια και να υπάρχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τη ρύθμιση για τα μυστικά καρτέλ. Οπότε, εξασφαλίσαμε ότι να έχει πρόγραμμα επί κάθε χώρα. Να υπάρχει μείωση ποινών και αμνηστία. Επίση να υπάρχει ομοιόμορφη εφαρμογή για όλα τα κρατημέλη και έτσι πετυχαίνουμε την ισορροπία μεταξύ του να υπάρχουν τα κίνητρα να ζητεί την ε, επίκαια μια εταιρεία και από την άλλη μεριά και την άλλη να υπάρχουν οι σχετικέ παροχές. Νομίζω ότι η ευελιξία που θέλουμε να προσδώσουμε στα μέτρα μας είναι κάτι που ενθουσιάσει όλους. Οι εθνικές αρχές να έχουν αρμοδιότητα ίσπραξη των χρηματικών ποινών και εν κατακλείδη όπως προαναφέρθηκε είναι πολύ σημαντική η πρόταση αυτή για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ήταν πιο στεγανούς τους κανόνες του ανταγωνισμού και ευπρόσδεκτες προτάσεις σας για βελτίωση των δικών μας. Να κινηθούμε ταχαίως και, και εσείς το είπατε αυτό και μπράβο σας και ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε τώρα να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Τι λέτε κύριε Σιγητά για δευτερολογία σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν μου, αν μου πείτε να, μιλήσε, να μιλήσω σύντομα, να μην απαντήσω σε όλες τις εμέρους παρατηρήσεις των συναδέλφων, απλά να τους ευχαριστήσω για το πνεύμα καλής συνεργασίας και στον κύριο Γκίκολ να ευχηθώ ε, χρόνια πολλά στον κύριο Ράιμοντ που δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα. Ίσως γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να είναι παρόν. Όπως και να έχει, νομίζω ότι τα βασικά θέματα έχουν εξεταστεί από τις διάφορες πλευρές και το τελικό θέμα θα είναι πώς θα βρούμε τη σωστή ισορροπία. Ακόμα και ο κύριος Γκίγκολτ ε, τόνισε στο τέλος ότι θα πρέπει να σεβαστούμε την αρχή του κράτους δικαίου. Αυτό θα πρέπει να το πετύχουμε έχοντας από την άλλη μεριά και ευελιξία. Πρόσεξα επίση αυτό που είπε ο κύριος Ντεκάιζερ. Ε, πιστεύουμε ότι είναι καλή η πρόταση, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία, ίσως να μπορέσουμε να τη βελτιώσουμε κάπως την πρόταση αυτή. Ε, και το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε όλες τις προτάσεις των συναδέλφων χωρίς να καταστρέψουμε συστήματα που λειτουργούν πολύ καλά. Θέλουμε να διορθώσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, απ' την άλλη δεν θέλουμε να αγγίξουμε τα συστήματα που λειτουργούν καλά. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί αυτή η ισορροπία. Και γι' αυτό επρόκειτο για κεντρική πρόταση ε, και ο κύριος Γκίγκολα αναφέρθηκε στην ε, κληρονομιά μας, ε, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο κύριος Σταρμπάτη. Ας προχωρήσουμε λοιπόν σε επικοδομητική συζήτηση. Ελπίζω να μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να κατέχει την πολύ καλή θέση που κατέχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να σας θυμίσω το χρονοδιάγραμμα. Ένα λεπτό, λάθος χαρτί διαβάζω. Παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης 9 Οκτωβρίου, προθεσμία για την ε, υπολογή τροπολογιών 20 20 Οκτωβρίου, 20 ε, Νοεμβρίου ε, συζήτηση και 4 Δεκεμβρίου ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας ε, διάταξη. Γενικό Προπολογισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 όλα τα τμήματα. Συντάκτης νομοδότηση, ο Μάρκο Φέρμπερ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι δεν είναι το πιο αγαπημένο θέμα της ε, ΕΚΟΝ αυτό, γι' αυτό πάντα κολλάμε στο Προεδρείο. Ε, έχουμε λοιπόν όλα τα τμήματα του προϋπολογισμού του επόμενου έτους. Έχουμε πάντα τις ε, τρεις αρχές, την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και οι αρχές αυτές ε, θα πρέπει να περικοδοτηθούν ανάλογα. Ε, έχω συναντηθεί και με τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές ε, της ΕΣΑΣ Βλέπετε λοιπόν ότι και οι ίδιες αρχές ενδιαφέρονται πολύ για την συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Έχω συγκρίνει τα, τις δομές των τριών ε, αρχών ε, και 112 θέσεις πλήρους απασχόλησης ε, προβλέπουμε για το επόμενο έτος. Αυτό είναι κάτι που συμφωνήσαμε το 2011 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Θα ήθελε δύο θέσεις παραπάνω από ό,τι προβλέπονται, διότι υπάρχουν διάφορα προγράμματα ψηφιακά τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν. Έχω εκπονήσει σχετικό κατάλογο και νομίζω ότι αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί. Θα ήθελα όμως πολύ να ακούσω και τις παρατηρήσεις ε, των συναδέρφων. Η ΕΣΜΑ έχει 156 θέσεις απασχόλησης. Παρακαλώ, αν κλείσετε το μικρόφωνο, θα μπορέσω ε, να γίνω πιο εύκολα κατανοητός. 156 ε, θέσεις πλήρους απασχόλησης, έχει 7 θέσεις λιγότερες από ό,τι προβλεπόταν. Αυτό όμως συνδέεται με το γεγονός ότι λόγω των κανόνων χρηματοδότησης οι εθνικές αρχές ε, δεν ήταν διατεθειμένες ε, να δώσουν περισσότερα χρήματα στην ΕΣΜΑ και γι' αυτό μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι σε εποχές ε, περιορισμένου δυναμικού είναι σημαντικό οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να ε, ασχολούνται μόνο με τα καθήκοντα που προβλέπονται στις εντολές τους ε, και επίσης θα πρέπει να ασχοληθούμε με τη χρηματοδότηση των ε, τριών αυτών. Ξέρω ότι η αναθεώρηση είναι το κατάλληλο σημείο να γίνει αυτό, την οποία περιμένουμε, αλλά επιτρέψτε μου την παρατήρηση ότι χρήσιμο θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, Ε, να μετακυλήσουμε μέρος ε, της χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών ε, στις επιχειρήσεις, στους συμμετέχοντες στην αγορά. Και τέλος, λίγα λόγια για το Brexit και οι τρεις εποπτικές αρχές θα επηρεαστούν από το Brexit διότι το Brexit έχει συγκεκριμένε συνέπειες και για τις ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές αγορές. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν επαρκές δυναμικό, ε, ανθρώπινο, ε, μηχανογραφικό κλπ. Ε, οι αρχές αυτές. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, έχουμε την ιδιαίτερη ε, κατάσταση ότι μετά την εγκατάλειψη του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να παραμείνει στο Λονδίνο. Αυτό θα επιφέρει επιπλέον κόστος. Ε, το θέμα είναι ποιος θα καλύψει το κόστος αυτό. Εγώ ως ε, εισηγητής προτείνω το κόστος ε, να το καλύψει αυτό που φταίει. Δεν θα είχε προκύψει το κόστος αυτό ε, εάν δεν είχε εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να καλύψει το κόστος. Επίσης, η μεταφορά της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών θα ήταν και καλή αφορμή να σκεφτούμε περαιτέρω την δομή, μήπως θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε ε, χρήματα για τις ε, τρεις ευρωπαϊκές επαπτικές αρχές. Η ΕΣΜΑ στο Παρίσι, ανά τετραγωνικό και ανά μήνα, ε, πληρώνει 350 ευρώ και μισό η ΕΙΟΠΑ, ενώ στη Φραγκφούρτη η ΑΙΟΠΑ πληρώνει 29 ευρώ το το μήνα ανά τετραγωνικό. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το κόστος ενοικίου. Και εάν ε, εξετάσουμε τα ενίκια θα μπορέσουμε να κάνουμε εξοικονομήσεις. Αυτά από μένα ως εισηγήτη και με ενημερώνουν ότι μπορώ να προεδρεύσω και θα συνεχίσω στα αγγλικά και δίνω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές και ξεκινάμε από τον Όλε Λούντβιξον από το S&D. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Φέρπερ για σύντομη και ε, περιεκτική ε, γνωμοδότηση. Αναφέρεται ε, στις ε, τρεις ε, αρχές, το EBA, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την ΕΣΜΑ και την ΕΙΟΠΑ. Ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών είναι αποφασιστική σημασίας στην σωστή εφαρμογή του δικαίου και για την διασφάλιση της σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης για να προωθήσουμε καλύτερα ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές θα ήθελα να τονίσω τη σημασία οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές ε, να ε, περιορίζονται στα καθήκοντα που ε, ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Για παράδειγμα, πρέπει να ασχοληθούν με τα τεχνικά πρότυπα εάν το επιπλέον δυναμικό θα μπορέσει να βοηθήσει τις ε, εθνικές αρχές να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, ε, τότε αυτό θα είναι χρήσιμο. Όσον αφορά τη μεταφορά τη ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών από το Λονδίνο, συμφωνώ και συμφωνώ ότι το επιπλέον κόστος θα πρέπει να το φέρει το Ηνωμένο Βασίλειο. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν παράλογο κατά τη γνώμη μου. Ε, διότι θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις των συμφωνιών. Θα υποβάλουμε ε, τροπολογία στην ε, γνωμοδότηση και ελπίζω να έχουμε καλή συνεργασία και να καταλήξουμε σε καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ όλα για το, την ομάδα ECR, ο καθηγητής Σταμπάτη στη θέση του κύριου Λούντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης. Ε, Μιλάω στο, στη θέση του σκιώδου συγητού από την ομάδα μας που δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα μεταξύ μας. Χαίρομαι λέγοντας ότι συμφωνώ με τα περισσότερα τα οποία πρότεινε ο εισηγητής ε, σχετικά με τις διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις ε, στην δημοσιονομική πολιτική. Επίσης, για τον φόρτο εργασίας των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι ο φόρτος αυτός περνάει από νομοθετικό έργο ε, σε σύγκληση και ε, ε, θα, πρέπει να αλλάξει λοιπόν κάτι. Επίσης εκτιμούμε ότι αναφέρεται την δυνατότητα εισαγωγής ορισμένων συνδρομών των συμμετεχόντων. Αυτό δεν φαίνεται καλή ιδέα να κόψουμε τον χρηματοδοτικό ρόλο των αρμοδίων εθνικών αρχών. Ε, για να είμαστε πιο πλήρεις, θα ήθελαμε να ε, ε, προσθέσουμε κάτι σχετικά με τον ρόλο των Ευρωπαϊκών Υποπτικών Αρχών ε, στην επίτευξη της σύγκλησης. Σχετικά με την ΕΣΜΑ και την ΕΟΠΑ θα ήθελα να προτείνω μια άλλη προσέγγιση από αυτήν που χρησιμοποιεί ο εισηγητής. Αντί να αναφερόμεθα σε συγχώνευση ε, οργανισμών που αυτό θα είναι μια πολιτική απόφαση νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να αναφερθούμε ε, στα κριτήρια αποτελεσματικότητας. Αυτό κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να είναι ένα κεντρικό κριτήριο στην λήψη αποφάσεων σχετικά ε, με την μεταφορά της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Υπάρχει ακυρτό περιθώριο ερμηνείας σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την εργασία σας και ελπίζω να ε, οριστικοποιήσουμε αυτήν τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ε, επίσης, ε, χαιρετισμού στον κύριο Λούντς, δεν βλέπω κάποιον από την ομάδα Άλντε που να θέλει να λάβει το λόγο. Όχι, δεν εγγραφήκατε. Από την Γκουε, Μιγγέλ, Μιγκέλ. Μιγκέλ, έχει το λόγο. Καλημέρα σας. Διαβάσαμε το κείμενο. Εκεί τη φαίνονται σημαντικά ζητήματα. Συμφωνούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος αυτών των αρχών. Πρέπει οι αρχές να έχουν τους πόρους που χρειάζονται, ούτως ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να είναι και αποτελεσματικές. Όσον αφορά τώρα την χρηματοδότηση, έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. Πρώτα πρώτα για τη συγχρηματοδότηση συμφωνούμε, αλλά είναι πάρα πολύ βασικό το να είναι ανεξάρτητες αυτές οι αρχές. Θα είναι δημόσιες και θα πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία όσον αφορά τις αρχές που ελέγχουν τις άλλες με τη σειρά τους. Οπότε θα πρέπει η Επιτροπή, η δική μας Επιτροπή, να καταλήξει σε ένα κείμενο με κριτικό πνεύμα. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο ύψος των περιστάσεων. Χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις, χρειάζονται, ε, ε, χρειάζονται ενέργειες που να δώσουν μια όθεση στην ε, οικονομία. Να δούμε τι μπορεί να γίνει με μέτρα όπως ε, μέτρα σχετιζόμενα με τα επιτόκια. Έχουμε την προσθετικότητα, έχουμε το πλάνο Γιούγκερ. Ε, χρειαζόμαστε και μια πολιτική συνοχής, η οποία να ανταποκρίνεται στο ύψο των περιστάσεων, διότι σήμερα η πολιτική αυτή έχει κάπως ατονίσει να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των πλουσιωτέρων και των λιγότερο πλουσιών χωρών. Έχουμε τις περιφερειακές χώρες της Ευρώπης που είναι φτωχότερες, αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά προβλήματα γιατί συμμετέχουν στην ΟΝΕ. Είναι σημαντικό, θεωρώ από πλευράς μακροοικονομικής, να υπάρχει ένας προϋπολογισμός πιο θαραλέως και με κατάλληλες επενδύσεις να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που τώρα πλήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Ο κύριος Γκίγκολ για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί γενικά συμφωνούμε με τις προτάσεις για τον προπολογισμό. Συμφωνούμε γενικά με τα όσα έκανε ο εισηγητής. Συμφωνούμε και με τα αξιόλογα στοιχεία που μας είπατε. Και για τα ενίκια έχετε δίκιο. Να μην χρησιμοποιήσουμε τη γνωμοδότηση αυτή για να συζητήσουμε φόλες της ύλης, γιατί δεν βγάζει πουθενά ε, μια τέτοια διαδικασία. Αυτά είναι για την Επιτροπή Προπολογισμού και για την Ολομέλεια. Θα υπάρξουν πολλέ απόψει για το πώ μπορεί να αλλάξει ο προπολογισμό, αλλά εμά δεν μα ωφελεί τέτοια κουβέντα. Οπότε θέλω επίση να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στη δουλειά μας το έργο της ε, Eurostat. Υπάρχει ε, πρόταση νομοθετική επ' αυτού. Πρόκειται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Μίλησαμε με την Eurostat στο Λουξεμβούργο. Τους δείξαμε γιατί είναι δυσλειτουργικό το website τους. Είναι δύσκολα τα δεδομένα τους. Υποσχέθηκαν να κοιτάξουν το θέμα και ίσως θυμάται και ο εισηγητής ότι ε, αυτά με την γιούσα τα έχουμε πει σχετικά με το πόσο εύχεστα πρέπει να τα δεδομένα τα έχουμε ξαναπεί, έχουμε δαπανίσει τόσα χρήματα, αλλά δεν μπορεί ο κόσμος να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα. Οπότε τέλος πάντων ε, ε, η καινούργια διεύθυνση της υπηρεσίας υποσχέθηκε και πάλι να βοηθήσει. Δεσμεύθηκε προς τούτο. Τώρα όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, θεωρώ ότι και αυτές θα πρέπει να διαθέσουν περισσότερους πόρους για προστασία των καταναλωτών. Αυτή είναι η εντολή τους άλλωστε. Και αν κανείς συγκρίνει το τι κάνει η ΕΠΑ ή ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτό το μέτωπο, ε, μπορούμε να προσπαθήσουμε περισσότερο. Δεν συμφωνούμε με την ε, παρατήρηση στο σημείο 2 του σχεδίου κειμένου. Εκεί αναφέρεται ότι αυτές οι υποπτικές αρχές θα πρέπει να διευρύνουν την εντολή τους. Εμεί θεωρούμε ότι αυτές οι αρχές ανέκαθεν κινούνται στα πλαίσια των αρμοδιωτήτων τους και ό,τι κάνουν καλύπτεται από την ευρεία εντολή που έχουν στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας πλαίσια. Επίσης, έχουμε αυτό το πρότυπο που αναφέρει στο σημείο 7, Twin Peak, και όπως έχει σήμερα η συγκυρία ίσως είναι η καλύτερη λύση. Βέβαια, απ' την άλλη δεν είμαι σίγουρος εάν τέτοια θέματα θα πρέπει να μπαίνουν σε τέτοιες γνωμοδίες για τον προπολογισμό. Δεν πρέπει να συζητήσουμε ε, το, το, τις, τις Επιτροπής για τις ε, υπηρεσίες τις Και μετά. Και, και έτσι να ολοκληρώσουμε το θέμα. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, υπερβάνς. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε εισηγητά. Βεβαίως πρέπει κάποιος να ασχοληθεί με τον προϋπολογισμό. Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Βεβαίως όταν βλέπουμε τους προϋπολογισμούς που διαχειρίζεται η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Βεβαίως, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές είναι ένα θέμα προτεραιότητας, αλλά όλοι ξέρουμε ότι γίνεται μια αναθεώρηση για αυτές τις υπηρεσίες και οργανισμούς και δεν μπορούμε ίσως με την γνωμοδότηση απλώς ε, δεν ξέρω αν θα συμμεριστεί ο εισηγητής στην άποψη αυτή, δεν μπορούμε εμείς να προκαταλάβουμε τη συζήτηση που θα λάβει η χώρα κατά την εξέταση των προτάσεων ε, που θα μας παρουσιάσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και από την άποψη αυτή νομίζω ότι το να θέλουμε να δώσουμε επαρκείς πόρους ε, στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές για να μπορούν να εκτελέσουν καλά τις υποχρεώσεις τους. Βεβαίως είναι κάτι καλό, δεν αντιτίθεμε ε, να υπάρξει μια χρηματοδότηση από τους ενδιαφερόμενους της αγοράς. Πρέπει να αφήσουμε ανοιχτές τις θύρες ε, ανάλογα με τη συζήτηση που θα έχουμε αργότερα. Αναφέρατε ένα είδος πλέγματος ανάλυσης ανάλογα με το επίπεδο των ο καθένας διαλέγει τα κριτήρια που του αρμόζουν ή που τον ενδιαφέρουν. Εγώ προτείνω να ξανακάνουμε έναν έλεγχο της, ε, το, της δομής ε, της ε, έδρας της Φραγκφόρτης της, της τράπεζας και να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής, αυτών των αγορών της οικοδόμησης στην ε, μεταφορά, με την εγκατάσταση των οργανισμών, ένα σημαντικό πράγμα είναι ότι όταν η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα ε, μετακομίσει από το Λονδίνο θα πρέπει να έχει για τα στελέχη την ίδια, το ίδιο επίπεδο γιατί δεν μπορούμε να μειώσουμε την ποιότητα των στελεχών ε, της ΕΜΠΑ επειδή θα γίνει μετακόμιση θα πρέπει δεν το λέω για να υποστηρίξω μια πόλη, αλλά ε, τα κριτήρια βεβαίως και το ενίκιο είναι ένα θέμα δημοσιονομικό σημαντικό, αλλά δεν είναι το μόνο κριτήριο, το καθοριστικό κριτήριο σε σχέση με τις, ε, τους άλλους τομείς που καλύπτονται, τα άλλα τμήματα που καλύπτει ο προϋπολογισμός με τον κύριο Στολαγιάν. Νομίζω ότι αποδώσαμε ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί την ε, και τη ΦΡΑΓ και την ΙΑΣΒ και νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε ε, στο θέμα αυτό και να χρησιμοποιήσουμε ε, την έκθεσή μας για να ελέγξουμε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις που κάναμε ε, στην έκθεση στο Λαγιάν και το θέμα των στατιστικών αναφέρθηκε θα ήθελα και εγώ να αναφέρω μια ανησυχία σχετικά με την μείωση των πόρων και των εργαλείων που τίθενται στη διάθεση των μονάδων που και ε, ε, καταπολεμούν ε, την διαφθορά και την βέλτιστη χρησιμοποίηση των μέσων απομείωσης της φορολογίας. Θα ήθελα να ληφθούν υπόψη και αυτά τα κριτήρια. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κανέναν άλλον να ζητά τον λόγο. Ε, ζητώ ε, να απαντήσει ο εισηγητής. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους. Υπάρχουν θέματα τα οποία έχουμε αποφασίσει σε διάφορα πλαίσια. Η βασική γραμμή ακολουθεί δηλαδή αυτά που έχουμε αποφασίσει τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά τα ενίκια, ήθελα να δείξω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Ε, δεν ήθελα να αμφισβητήσω τις έδρες ε, των ε, οργανισμών αυτών. Ξέρω ότι στο Παρίσι υπάρχουν κτίρια με χαμηλότερα ενίκια και επίσης ο οργανισμός βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο. Απλά ήθελα να πω ότι υπάρχουν και άλλα κτίρια στο Παρίσι με χαμηλότερα ενίκια, τα οποία όμως είναι αρκετά ε, καλά. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις πολλές παρατηρήσεις. Όσον αφορά τις στατιστικές, ε, σίγουρα θα μπορέσουμε να το συμπεριλάβουμε και αυτό. Κατά τα άλλα, θα εξαρτηθούν ε, όλα από το τι θα κάνει η Επιτροπή Προϋπολογισμού τελικά ε, με την απέραντη σοφία της. Ε, έχουμε δει και άλλες φορές οι συμβιβασμοί που με πολύ κόπο εκπονήσαμε τελικά να συμπεριλαμβάνονται στην τελική πρόταση. Θα συνεχίσω στα αγγλικά τώρα, πρωτού να ε, ξαναδώσω την Προεδρία στον Πρόεδρο. Ε, 20 Ιουλίου στις 10 είναι η προθέσμια την κατάθεση τροπολογιών και ο εισηγητής ε, θέλει στις 29 Αυγούστου ε, να οργανώσει συνάντηση σκιωδών, διότι στις 30 θα έχουμε την εξέταση και ψήφιση της, ε, των τροπολογιών. Ξέρω ότι είναι η εβδομάδα που όλοι επιστρέφουμε από τις διακοπές μας και που ξεκινάει Τετάρτη για μας τα μέλη της ΕΚΟΝ, αλλά θα εκτιμούσα εάν Τρίτη βράδυ ή αργά το απόγευμα θα μπορούσαμε να έχουμε συνάντηση των σκιωδών για να προετοιμάσουμε τις ψηφοφορίες. Ειλικρινά, δεν βλέπω να υπάρχει άλλη δυνατότητα. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι στις 19. Πρέπει να ψηφίσουμε Παρακαλώ οι σκιώδεις να περιμένουν δηλαδή πρόσκληση από τον εισηγητή για συνάντηση των σκιωδών ε, στις 29 Αυγούστου το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, παραδίδω την Προεδρία στον Πρόεδρο. Ευχαριστώ Μάρκους. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Δεν βλέπω όμως να είναι παρόν ο εισηγητής. Έχει ένα κείμενο εκεί. Ε. So we need Πρέπει να περιμένουμε τον κύριο Σίμων, λοιπόν. Εκτός αν κάποιος σκιώδης θέλει να πάρει τη θέση του. Welcome. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίζω τον εισηγητή. Όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε στο σημείο 8. Εξετάζουμε τις τροπολογίες, θα έχουμε μετά την ψηφοφορία. Ευχαριστώ τον εισηγητή και όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την καλή τους εργασία που μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε ταχύτατα αυτό το μικρό μέρος του τραπεζικού πακέτου για να έχουμε καταλήξει πριν από το τέλος του χρόνου. Ο εισηγητής έχει καταθέσει συμβιβαστικές τροπολογίες. Σας δίνω τον λόγο για να παρουσιάσετε αυτές τις τροπολογίες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την επικοδομητική συζήτηση που είχαμε στο πλαίσιο των σκιωδών εισηγητών. Ε, καταφέραμε να καταλήξουμε σε τέσσερις συμβαστικές τροπολογίες ε, που ε, συνοψίζουν αυτά που επιθυμεί μια μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Mm. σε κάποια άλλα σημεία δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμβασμό. Σημαντικό όμως είναι για μένα ότι από τις 185 τροπολογίες που λάβαμε, που είναι πάρα πολλέ, πάνω από τις 60 ε, είναι απαράδεκτες διότι δεν αναφέρονται στο τμήμα που ψηφίζουμε τώρα, αλλά ε, στο, ε, στη διαδικασία που θα ακολουθήσει. έχουν συμπεριληφθεί στις ε, συμβιβαστικές ε, τροπολογίες ε, όλες οι υπόλοιπες σε, κάποια, σε περίπτωση που κάποια από τις συμβιβαστικές ε, καταψηφιστεί θα πρέπει να τις ψηφίσουμε μία προς μία και θα πρέπει να θεωρηθούν απαράδεκτες. Όσον αφορά λοιπόν το IFRS 9, το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9. Ε, Θέλουμε περισσότερη σταθερότητα, περισσότερη ασφάλεια. Οι πράσινοι και οι γκουε ε, θέλησαν κρατική προσέγγιση και για λόγους ασφαλείας ε, και επειδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει μια τέτοια προσέγγιση. Το κάνει όμως αυτό επειδή θέλει να απλοποιήσει την ζωή των οικονομικών φορέων. Αλλά οι οικονομικοί φορείς λένε ότι δεν χρειάζεται απλούστευση στον τομέα αυτών. Και τελικά τι είναι πιο ασφαλές, ε, κρατική ε, προσέγγιση που δεν θα μπορέσει να μια στατική προσέγγιση που ναι, να μην μπορεί να διορθωθεί εκ των υστέρων ή να έχουμε μια δυναμική προσέγγιση. Θα θέλαμε ε, δυναμική προσέγγιση κάθε χρόνο να μπορέσουμε να κάνουμε τροποποίηση των ε, προϋποθέσεων. Διότι βλέπετε πόσο γρήγορα αλλάζει ο κόσμος, πόσο γρήγορα μπορεί να στραφεί από τα αριστερά στα δεξιά και από το ε, καλό στο κακό. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε δυναμική προσέγγιση, όχι στατική. Ε, έχουμε κάποιε επιφυλάξει ε, σχετικά με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύουμε ότι είναι υπερβολικά γενναιόδορη απέναντι στι τράπεζε. Και στην συμβαστική πρόταση λέμε ότι μπορούμε να εμποδίσουμε οι βέβαιες ζήμιες να μην εξαφανιστούν ε, σε μια ποσόστοση δύο κεφαλαίου. Επιπλέον ε, έχουμε εδώ ένα στοιχείο που ε, διασφαλίζει οι ζημιές που έχει υποστεί κανείς που δεν έχουν ε, αναφερθεί να μην μπορούν να λαμβάνονται υπόψη. Γιατί τι ζημίες μιλάμε. Μιλάμε για ζημίες που στο παλιό πρότυπο 39 έχουν διαπιστωθεί, δεν έχουν αναφερθεί όμως. Οι ζημιές που, έχουν, που έχει ήδη υποστεί κανείς να μην μπορούν να εξοραϊστούν στον υπολογισμό. Άλλο σημαντικό θέμα εδώ είναι ότι θέλουμε να αποφύγουμε την προτίμηση τραπεζών ε, που να χρησιμοποιούν εσωτερικό μοντέλο. Ήδη πριν από την εφαρμογή του Δύχ 9 η έκθεσή μας ε, με τις, ε, με τις συμβαστικές τροπολογίες δείχνει ότι όταν υπάρχει κέρδος ε, που να ξεπερνάει την ζημία αυτό μπορεί να προσθεθεί στο κεντρικό κεφάλαιο. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει πενταετή μεταβατική φάση ε, με προοδευτική μείωση, δηλαδή στο πρώτο έτος να προβλέπεται ε, απόλυτη ουδετερότητα. Οι τροπολογίες που λάβαμε πηγαίνουν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ε, πολλοί θέλανε ε, συντελεστεί ένα όσον αφορά την ουδετερότητα για ένα έτος. Ε, μερικοί ήθελαν για δύο χρόνια, άλλοι δεν ήθελαν καθόλου συντολιστεί ένα, αλλά πολύ χαμηλότερο. Η συμβαστική πρόταση προβλέπει το πρώτο έτος συντελεστεί 1,9 δεύτερο έτος 0,8, τρίτο έτος 0,6, 0,4 το τέταρτο έτος και τέλος 0,2 το πέμπτο έτος, ώστε ήδη από την αρχή να μην έχουμε απόλυτη ουδετερότητα, 0,9 το πρώτο έτος ως τελεστή, συγγνώμη, Και έτσι έχουμε διατηρήσει το μεταβατικό διάστημα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, αλλά έχουμε ε, αυξήσει κάπως την ουδετερότητα. Νέο επίσης είναι η αρχή ότι οι τράπεζες ήδη πριν τη μεταβατική περίοδο ε, έχουν επιλογή αν θέλουν να εκμεταλλευτούν το σύνολο της μεταβατικής περίοδου ή μήπως δεν θέλουν καθόλου μεταβατική περίοδο. Η μόνη εξαίρεση προβλέπεται για τράπεζες που το πρώτο έτος αποφασίζουν ότι θέλουν μεταβατική περίοδο. Με την συμφωνία της εποπτικής αρχής οι τράπεζες αυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, το ίδιο σύστημα για τα έτη 2 έως 5. Έτσι μπορούν οι τράπεζες ε, να προσπαθήσουν ε, να ε, μην έχουν μεταβατική περίοδο, αλλά σε περίπτωση που απετύχουν το δεύτερο έτος να περάσουν στη μεταβατική ρύθμιση. Κατόπιν έχουμε τροπολογίε τροπολογίες των συναδέλφων Κάρας και Φαν Ιουγενόη που έχει να κάνει με την εντολή της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Το θέμα είναι λοιπόν ο συντελεστής μόχλευσης ε, πώς θα αναφέρεται στην περίπτωση όπου εφαρμόζεται η μεταβατική περίοδος και σε φάσεις όπου δεν εφαρμόζεται. Κατόπιν ε, έχουμε τα μεγάλα ανοίγματα. Αυτό το βλέπετε στην συμβιβαστική β. Έχουμε λοιπόν ε, εδώ ρυθμίσεις ε, για ε, δάνεια σε ε, ξένο νόμισμα. Και από την 1η Ιανουαρίου 2018 θα πρέπει να ισχύουν οι κανόνες και κάτι που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να οδηγήσει κάποια κράτη-μέλη σε μεγάλα προβλήματα. Ε, εμείς έχουμε λοιπόν εδώ μία τριετή μεταβατική φάση, 100% του κεφαλαίου το πρώτο έτος, 75% το δεύτερο και 50% το τρίτο. Ε, έτσι μπορούμε να αποφύγουμε αυτά τα, ε, τα πολύ απότομα αποτελέσματα. Λόγω της λάθους αναφοράς στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση. Οι τροπολογίες αυτές έχουν αποτελέσει αντικείμενο συνεννόησης με το Συμβούλιο και ε, τα δάνεια που είναι εκπεφρασμένα σε ξένο νόμισμα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αποκλείονται από την ε, ρύθμιση. Ενώ εμείς λέμε ότι όλα τα κρατικά δάνεια σε ξένο νόμισμα συμπεριλαμβάνονται. Όλοι δηλαδή καλύπτονται από την μεταβατική ρύθμιση. Πιστεύω λοιπόν ότι και εδώ όσον αφορά τα μεγάλα ανοίγματα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες. Ευχαριστούμε κύριε Σίγητα. Πάρα πολύ εύστοχοι η οι με του κλείσατε και τώρα για το ΕΛΚ. Ο σκέδος ο κύριος Κάρας. Κύριε Πρόεδρε. Και εκ μέρου του ΕΛΚ μπορώ να πω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις συμβιβαστικέ τροπολογίες, διότι πιστεύουμε ότι αποτελούν μια πολύ καλή μέση οδό. Από τη μία θέλουμε δυναμική προσέγγιση, που να συμπληρώνεται από ένα στατικό στοιχείο, κάτι που ανταποκρίνεται στα πρότυπα της Βασιλείας. Έτσι, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα έχουν αρκετό χρόνο για να ετοιμαστούν όσον αφορά τα μεγάλα ανοίγματα. Η πενταετής μεταβατική περίοδος ε, συμμορφώνεται και με τις ε, διατάξεις της Βασιλείας. Το ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να αποφασίσουν αν θέλουν βαθμία εισαγωγή ή όχι, νομίζω ότι ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης, ε, συμφωνούμε που έχουν συμπεριληφθεί οι κατευθυντήριες γραμμές ε, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής σχετικά με την υποβολή αναφορών. Και στηρίζουμε και στην παράγραφο 3β την κλιμακωτή προσέγγιση. Επίσης επικροτώ το ότι ο εισηγητής έχει συμπεριλάβει το κείμενο του Συμβουλίου όσον αφορά την βαθμία εισαγωγή, όπου το πεδίο εφαρμογή είναι κάπως πιο στενό. Άλλωστε δεν μιλάμε εδώ για νέα κατηγορία ανοιγμάτων, μιλάμε απλά για μια πολύ σωστή κατηγοριοποίηση. Καλό λοιπόν τους ε, συναδέρφους μου από το ΕΛ και να υπερψηφίσουν τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες ε, που έχουν συμπεριλάβει όλες τις τροπολογίες μας. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Κοραφανή εκτός αν θέλει η κυρία Σαμπάτη εξ ονόματος του κυρίου Φόξ να λάβει το λόγο. Ναι, θα μιλήσω εξ ονόματος του κύριου Φόξ. Ναι, συγχαίρομαι τον εισηγητή για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του φακέλου. Η ECR υποστηρίζει τις ε, συμβιβαστικέ τροπολογίες και τη δυναμική προσέγγιση, διότι νομίζω ότι είναι η καλύτερη μέθοδος και πιο αποτελεσματική Ο στόχος είναι οι τράπεζες να έχουν καλή κεφαλαιοποίηση χωρίς να μειώνουν το δανεισμό στην πραγματική οικονομία. Οι ρυθμιστές θα πρέπει να δουν ε, ποιες ε, είναι τα αποτελέσματα του νέου IFRS και πώς ε, να ανταποκριθούμε στις περιστάσεις. Έχουμε ε, εισαγάγει ορισμένες ε, τροπολογίες για την ε, μεταβατική περίοδο, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι με τις συμβιβαστικές τροπολογίες και θα θέλουμε να αρχίσουμε την, το διάλογο για διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κόρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για την αγορά και την πραγματική οικονομία ε, ταχυρύθμως να προωθήσουμε αυτή την νομοθεσία και νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε αυτό το συνέστημα ότι είναι κατεπήγον το θέμα και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή ε, για τις ε, προτινόμενες συμβιβαστικές τροπολογίες. Έκανε πολύ καλή εργασία για να ε, ε, εγκρίνει πολλές τροπολογίες από όλους μας και αυτό αντανακλά ε, την ικανοποίηση ώστε να γίνουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες πιο ασφαλείς και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον τομέα των επιχειρήσεων. Επίσης είναι σημαντικό οι τράπεζες να εφαρμόσουν το συντομότερο δυνατόν τους νέους κανόνες του ΔΠΧΑ νέα και επίσης θα πρέπει να παρακολουθούμε να υπάρχουν ίσοι όροι, ίσοι όροι λειτουργίας ε, για την μεταβατική περίοδο ούτως ώστε μικρά τμήματα του α 9 να εφαρμοστούν και μετά θα υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής. Είμαι ευτυχής που υπάρχει τώρα δυνατότητα η πιο φιλόδοξη ε, βεβαίως να έχουν την ε, ευκαιρία να αλλάξουν, ελπίζω, και επίσης υιοθετώ την επιλογή σας για την δυναμική προσέγγιση η οποία τώρα προτείνεται εφόσον αυτή η προσέγγιση προσαρμόζεται καλύτερα στο περιτορινό περιβάλλον και λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους ε, του συστήματος. Ίσως το θέμα είναι λίγο πιο περίπλοκο αλλά αυτοί που θα εργαστούν με αυτό το σύστημα, αν δεν πιστεύουν ότι είναι πρόβλημα, γιατί εμείς να θεωρούμε ότι είναι πρόβλημα. Ε, κλείνω λέγοντας ότι υποστηρίζω τις συμβιβαστικές τροπολογίες, διότι νομίζω ότι επιφέρουν μια σωστή ισορροπία ε, και περιμένω ότι θα συνεργαστούμε καλά ε, και στο μέλλον. Ναι. για την ΚΟΕ, ο Φάβιο, για την ΚΟΕ. Ναι. Θα ήθελα να λάβω τον λόγο εξ ονόματος του κάτι που δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την εργασία του και την εκποδομητική ε, συζήτηση. Βεβαίως ε, δεν δεν ζητούμε τίποτα το ακραίο εμείς ε, θέλουμε την, ε, την κατάλληλη ε, ενιαία εποπτεία και τον μηχανισμό. Δεν θέλουμε στατική προσέγγιση, θέλουμε δυναμική και για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τους συμβιβασμούς, διότι νομίζω ο η στατική προσέγγιση για ορίζοντα τριών ετών θα ήταν πολύ καλύτερη και λυπούμεθα που η Κομισιό δεν, δεν δέχεται οι τράπεζες να μπορούν να απομακρυνθούν αφού υιοθετηθεί το ΔΠΧΑ9 νομίζουμε ότι θα πρέπει να ακούσουμε καλύτερα τις εποπτικές αρχές και να είμαστε πολύ πιο ε, προσεκτικοί. Υπάρχουν πάρα πολλέ για να μην υπάρξουν εκ, από την αρχή αδυναμίες. Ευχαριστώ, Σβεν Γκίγκολτ. Πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς ε, την επαγγελματική εργασία, ε, το, για την επαγγελματική του εργασία των εισηγητή που πόρεσε αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει το θέμα δεν θα πρέπει το πρώτο έτος να υπάρχει πλήρες offsetting. Βεβαίως δεν συμμεριζόμαστε τη γνώμη της πλειοψηφίας, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει cliff effect problem, όλα αυτά τα προβλήματα είναι γνωστά εκ των προτέρων Νομίζουμε ότι, γιατί, ότι δεν υπάρχει ε, συνολική ισορροπία σε αυτήν την έκθεση με τα 3-5 χρόνια, όχι ε, στην, ε, στο κάτω άκρο της σειράς Βασιλείας. Θα θέλαμε μια συντομότερη περίοδο. Επίσης, συμφωνούμε ότι η δυναμική προσέγγιση ε, δεν ξέρω αν είναι καλύτερα. Θα προτιμούσαμε να ακολουθήσουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την EBA. και να συμπεριληφθεί εδώ ο χρηματοπιστωτικός τομέας και τέλος ελπίζουμε ότι όταν θα εργαστούμε μαζί για το τραπεζικό πακέτο στο σύνολό του θα επανέλθουμε σε μια ισορροπία που να μειώνει περισσότερο τον κίνδυνο παρά να υποστηρίζει εκ των υστέρων μετά από πολλά έτη συζητήσεων για τον ΔΠΧΑ9 όπου λέμε ότι δεν είναι τέλειοι οι κανόνες αλλά ότι είναι πιο προσεκτικοί να μην επανέλθουμε τότε ε, σε έναν τρόπο όπου το κοινοβούλιο αυτό θα ζητήσει ε, οι κίνδυνοι που παραμένουν στον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο να πρέπει πιο αποτελεσματικά να αντιμετωπιστούν. Νομίζουμε ότι χρειάζεται μια ισορροπία με περισσότερη αναλογικότητα και αυτό πρέπει να πράξουμε και θα ήθελα επίσης να πω ότι επειδή ο εισηγητής αναφέρθηκε στο θέμα αυτό ότι υπάρχουν πολλά, πολλές απαράδεκτες ε, τροπολογίες και μόνο ε, για λόγους διαφάνειας προήλθαν από δύο ομάδες ε, που αποτελούνται από ευρωσκεπτικιστές. Και είναι καλό να ονομαστούν σαφώς αυτοί που χρησιμοποιούν αυτόν τον τεχνικό φάκελο για θέματα, για θέματα που είναι εκτός φακέλου αυτού. Ευχαριστώ. Ο κύριος ευχαριστώ πρόεδρε. Όσον αφορά το πώς θα εξασφαλίσουμε κάποιο είδου καλύτερη προσέγγιση από πολιτικής πλευράς για μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι τράπεζε να υποστηρίξουν το ΣΜΜΕ και τι οικογενειακέ επιχειρήσεις, αλλά να υπάρχει τέτοια προσέγγιση. Ε, αυτή τη φορά συμφορώ με τους προλαλήσαντε. όντω έτσι θα πρέπει να τεθούν κάποιε προποθέσει. Επίση, θα πρέπει αυτού του είδους ε, οι κεφαλικές ε, απαιτήσει να νομοθετηθούν ε, για τι τραπέζες που αναπτύσσουν τέτοιε δραστηριότητε. Θεωρούμε όσο δεν πρέπει να τις πολύ γιατί ήδη έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ <clears throat> από την σήμερα ισχύουσα τραπεζική εποπτεία άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ε, κρίση όσον αφορά τα χρηματοδοτικά προϊόντα, γιατί η κρίση ήδη χτύπησε πάρα πολύ τις ε, τράπεζες όσον αφορά τις πιστώσεις προς την ε, πραγματική οικονομία. Οπότε θα πρέπει να δούμε το ότι δυστυχώς δεν γίνεται να υποστηρίξουμε αυτό το κείμενο. Αλλά είναι δυναμική αυτή η προσέγγιση και εμείς θα ακολουθήσουμε μια προσέγγιση που θα βελτιώσει την πρόταση. Ευχαριστούμε κύριο Τζάνι. Ε, πάρα πολύ σύντομα. Ε, βέβαια και δεν συμφωνώ με αυτή τη νέα νομοθεσία. Θεωρώ ότι πρόκειται να επιφέρει πάρα πολλά προβλήματα παρά το ότι πρόκειται για κάποια απόπειρα ε, του να μας το θωρακίσει από τους κινδύνους του παρελθόντος σε σχέση με αυτή την καινούργια υιοθετηθής αρχή αφετηρία είναι λάθος. Εν προκειμένου θα πρέπει δηλαδή να δούμε πώς να έχουμε όσο γίνεται περισσότερη προστασία σε σχέση με υποτιμήσεις και με κρίσεις. Ε, είναι λάθος προσέγγιση αυτή. Το πρόβλημα των MPL κυρίως για την Ευρωζώνη δεν προκύπτει, δεν προκύπτει διότι είχαμε κάποιες ε, τοποθετήσεις που δεν ήταν πολύ προσεκτικές. Στο ΣΟΛ 24 ώρες έλεγε ένας αρθρογράφος ότι το πρόγραμμα αφορά, το πρώτο αφορά το αποτελέσματα της κρίσης, αυτά τα οποία αντιμετώπισε για πρώτη φορά η Ευρώπη και η Ευρωζώνη. Άρα ο μόνος τρόπος επίλυσης αυτού του προβλήματος είναι η οικονομική ανάπτυξη. Ε, αυτό με τέτοια νομοθεσία και με την νομοθεσία που Τώρα πέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται αυτά. Φρενάρουν την ανάπτυξη. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο. Δεν βλέπω να ζητεί κάποιο για το Κατσουδιάι. Άρα να δώσουμε το λόγο ξανά στον εισηγητή. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις εισηγητές ε, και για την επικοδομητική συζήτηση σήμερα και θα ήθελα ως διευκρίνηση να πω το εξής. Δεν διαφωνούμε σχετικά με το αν θέλουμε περισσότερη ασφάλεια και μείωση του κινδύνου ή όχι. Διότι κάπως έτσι φάνηκε. Το θέμα είναι πώς θα το πετύχουμε αυτό. Εκεί διαφωνούμε. Για παράδειγμα, εγώ νομίζω ότι ο κίνδυνος του cliff effect είναι μεγαλύτερος από ό,τι νομίζει ο συνάδελφος Γκίγκολτ. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε το εξή. Δεν υπάρχει κανείς εδώ που να, είναι, που να αμφισβητεί τη βασική πρόθεση αυτής της διαδικασίας ε, fast tracking, της συντομευμένης διαδικασίας που προτείνουμε. η πλειοψηφία όπως και τα περισσότερα κράτη-μέλη ε, στο Συμβούλιο πιστεύουν ε, ότι ε, μια δυναμική προσέγγιση θα ήταν καλύτερη. Εάν λοιπόν αύριο τα πράγματα πάνε ανάλογα με τη σημερινή συζήτηση θα καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα της ΕΚΟΝ. Ε, και ο συνάδελφο Κίκολ και ο συνάδελφο Μάζη μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη. Θα δούμε τελικά ποιο θα έχει δίκιο. Ευχαριστώ όλου πάντω για την καλή συνεργασία. Και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μα με εξίσου επικοδομητικό πνεύμα και με τις ε, διάφορες ε, διαφωνίες που υπάρχουν. Νομίζω όμως ότι το ξεκίνημα ήταν ήδη πολύ καλό. Και ήταν πολύ καλή και η συνεργασία σας. Ευχαριστώ θερμά. Grazie. Senza dubbio un buon inizio. Il voto avrà Ωραία, καλά ξεκίνησε αυτή η διαδρομή. Το και σε λίγο θα κάνουμε την ε, ψηφοφορία πάνω στο επόμενο σημείο, αλλά δεν βλέπω τον εισηγητή. Sì. You represent Mr. Eh, Α, θα μιλήσετε αντί του κυρίου Χόγμαρ. Πάμε τότε στην συζήτηση για το επόμενο θέμα. Να αποφασίσαμε να επιταχύνουμε όσον αφορά αυτή την κατάταξη χορογράφη. Αλλιώς τα είχαμε αποφασίσει στην αρχή, αλλά κατόπιν καταλήξαμε να επιταχύνουμε τη διαδρομή αυτού του θέματος. Οπότε δεν μπορώ να ευχαριστήσω τον τον κύριο Χόκμαρ που συνέταξε αυτό το κείμενο. Είναι ενθαρρυντικά τα όσα έκανε που έχει θεραμιστεί με τα όσα ήθελε και το Συμβουλίο. Και δίνουμε το λόγο στον κύριο Χάρας. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν είναι δυνατόν για τον κύριο Χόκμαρκ να είναι παρόν σήμερα, μου ζήτησε χθες ε, να διαβάσω την εξής δήλωση στο όνομά του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την δημιουργία μιας νέας κατηγορίας μη εξασφαλισμένων ε, χρεών για να ε, μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης. Ο κύριος Χέκμαρκ γενικά ε, συμφωνεί με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναγνωρίζει όμως ότι μπορεί να μην είναι πολύ εύκολο να επιτευχθεί αυτό σε μια σειρά κρατών μελών, όπου η ιεράρχηση ε, θεσπίζεται στην εθνική νομοθεσία. Για να πετύχουμε ασφάλεια δικαίου για τους ε, επενδυτές και εκδότες θα πρέπει να υπάρξουν επιπλέον ρυθμίσεις. Για το λόγο αυτό, ο κύριος Χέκμαρκ είναι κατά ενός καθεστώτος ε, που διασφαλίζει τις διατάξεις που έχουν ε, ε, θεσπιστεί πριν την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ελάχιστη διάρκεια οριμότητα ενό έτου διάρκεια λήξη. Ο κύριο Χόικμαρκ προτείνει να μην υπάρχουν εδώ ελάχιστε προποθέσει. Και αν τα μέσα αυτά έχουν ε, προθεσμία λήξης ε, χαμηλότερη, τότε δεν ε, θα ε, αντιστοιχούν στις απαιτήσει ε, ιδίων κεφαλαίων και αποδεκτών ε, υποχρεώσεων. Ο κύριος Χέκμαρκ δεν θέλει να αποκλείσει εκ των προτέρων κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δημιουργώντας νέα κατηγορία με ημερομηνία λήξης μικρότερη του ενός έτους. Επίσης, όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας ε, στο άρθρο 72 ε, του του ε, κανονισμού για τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις θα πρέπει να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή συνοχή μεταξύ των διαφορών νομοθετημάτων. Ο κ. Χόικμαρτ θα ήθελε τέλος να τονίσει ότι είναι σημαντικό για τους επενδυτές και εκδότες να υπάρξει σύντομα σαφήνεια σχετικά με την ιεράρχηση. Ο κύριος Χόδεκμακ προσβλέπει στην ε, συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές για να βρεθεί κοινή προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Κάρας. Η υπερβόνς περέσαν αντί του κύριου Περέιρα. Ε, ο συνάδελφος ε, αντιπροσώπησε τον ε, κύριο Χόκμαρ και εγώ τον Περίρα. Ευχαριστή τον συγητή και επίσης ευχαριστή για την προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος όσον αφορά την ε, πρωτοβουλία του Συμβουλίου με την ε, ταχεία διαδικασία. Πάντοτε οι σοσιαλιστές αυτό επιθυμούσαμε, οπότε χαιρόμαστε που συμφώνησε με τέτοια προσέγγιση ο συγητής του ΕΛΚ. Ακριβώς ε, όπως ε, προελέχθη θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση θα πρέπει να προωθηθεί. Θα πρέπει τα πράγματα να έχουν μια προβλέψιμη, ξεκάθαρη διαδρομή. Θα πρέπει να έχουμε ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις ε, αγορές. Και θα πρέπει το συντομότερο οι τράπεζες να μπορέσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις που τάσσονται εδώ. Το TLAC και το MREL. Και έτσι να συνάδουν τους με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Θα πρέπει ταχαίως να ενεργήσουμε. Και έτσι οι τράπεζες το συντομότερο δυνατόν να μπορέσουν να διεκπεριώσουν όσο γίνεται περισσότερες τέτοιες οφειλές και πτωχεύσεις. Επί της ουσίας έχουμε τρεις παρατηρήσεις και μία τέταρτη προσωπική δική μου. Θεωρούμε ότι η κατάργηση της ελάχιστης διαρκείας του ενός έτους δεν είναι καλή ιδέα. Έτσι. Θα υπήρχε διαφορά σχέση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΜΡΕΛ. Αυτό θα εγκυμώνει προβλήματα όσον αφορά την ε, αξιοπιστία των τραπεζών. Επίσης έχουμε και την ιδιωτικη παραγραφο παράγραφο 4α. Πώς θα διαχειριστεί κανείς την, ε, την οφειλή και ε, πώς θα γίνεται το λεγόμενο grandfathering της οφειλής. Αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί με κριτήρια επιλεξιμότητας και από πλευράς ΜΡΕΛ για τις προϋποθέσεις που τάσσονται και τις καθεντήρες γραμμές. Επίσης, αυτή η περίοδος 12 μηνών ως μεταβατική περίοδος. Είναι σημαντικό γιατί όλη αυτή η σύντομη διαδικασία fast track αποσκοπεί στο να μπορέσουν οι τράπεζες το συντομότερο δυνατόν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις διατάξεις. Τελευταίο τώρα που θέλω να προσθέσω είναι οι προϋποθέσεις που αφορούν τα embedded derivatives, τα embedded παράγωγα. Θα πρέπει αυτό το οποίο πρότεινε το Συμβούλιο να το, δούμε εμείς πώς το προσυγκινούμε και πώς θα ρυθμιστούν αυτού του είδους τα παράγωγα, τα embedded derivatives. Ο κ. Καμάλ για την ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και την και ευχαριστώ τον εισηγητή, τους σκιώδεις εισηγητές ε, Κύριε Μπέρες, ε, συμφωνώ με ορισμένα τα οποία είσατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον Γκούναρ Χεκμάρκ για την εργασία του και βεβαίως έχουμε προτεραιότητα για το θέμα αυτό και δεν ξέρω για την μεταφορά των κανόνων και θα θέλαμε να διευκρινίσουμε γενικά την απέτηση ΜΡΕΛ και δεν ξέρω ναι, σε σχέση με τα όσα είπε και η Ρεπέρες για τις ε, μεταβατικές ε, διατάξεις θα πρέπει να υπάρχει ε, κάποια σαφήνεια. Ένα πράγματα τα οποία Άκουσα, άκουσα τον κύριο Κάρας που αναφέρθηκε σε κάτι, αλλά θα ήθελα ε, να ε, σχετικά με την 9 και 20, σχετικά τις ε, διατάξεις για τις υποχρεώσεις για ένα έτος. Θα πρέπει για ορίμανση να υπάρχει κάτι που να συνάδει με παγκόσμια πρότυπα. Και νομίζω ότι το θέμα του ενός έτους σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνολικό επίπεδο, είναι σημαντικό ε, για την απορρόφηση των ζημιών. Σε αυτό το στάδιο θα ήμουν επιφυλακτικός με την πρόταση του εισηγητού, αλλά μπορούμε να έχουμε μια συζήτηση. ελπίζω ε, να, έχουν καλά λόμπι οι τράπεζες. Ε, θα ήθελα σαφήνεια για τους κανονισμούς των διαφόρων οντοτήτων των οικοδομικών και θα αναφέρει ότι θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη η διαδικασία. Τι, ε, τι εννοεί με αυτό, θα ήθελα περισσότερες ε, λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Βεβαίως, αυτή αποφασίσαμε να έχουμε δύο εκθέσεις ε, παράλληλες σχετικά με το θέμα αυτό διότι η ερμηνεία μου είναι άλλη. Υπάρχει η αναφορά αυτή σε αυτό το πακέτο, η προσέγγιση στο πακέτο με δύο ε, εκθέσεις, ούτως να υπάρχει κάποια συνεκτικότητα. Ο κύριος Κανασσός θα τον απαντήσει, ο κύριος Κορμιγέ για την ομάδα Άλντε, όχι. Όχι, σήμερα έχουμε πολλές αντικαταστάσεις. Ναι, στην ε, εγώ μιλάω για τον κύριο Κορνιγέ. Βεβαίως χαιρόμεθα που βλέπουμε ότι έχουμε το, την αρχή αυτή της ταχύρυθμης αντιμετώπισης, fast track, ο κύριος Κορνιγέ βεβαίως υποστηρίζει το σχέδιο έκθεση, αλλά έχουμε τις ίδιες επιφυλάξεις που ήδη ανέφεραν η Περβάνς και ο Σαΐντ σχετικά με τις τροπολογίες 20 και 23, δηλαδή η, ε, διαγραφή σχετικά με το λιγότερο του ενός έτους. Αυτό είναι προβληματικό εφόσον οι ε, πρώτης εξασφάλισης ε, προτιμόμενες ε, κατηγορίες σχετικά με τα δάνεια, τα βραχυπρόθεσμα που έχουν υψηλή ρευστότητα, ίσως η δυνατότητα της διάσωσης με ίδια μέσα, ίσως επιφέρει κάποιο κίνδυνο. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη συζήτηση. Αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φάβιο Ντεμάζη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τον κύριο Κάρας που παρουσίασε εδώ την εισήγηση. Βεβαίως την πρόθεση όλες οι υποχρεώσεις να είναι διασώσιμες με τα ίδια μέσα ε, και βεβαίως η κατηγορία των senior, των πρώτης προτεραιότητας, ε, θα πρέπει να είναι σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει, έχει μινιμαλιστική προσέγγιση σε σχέση με την ιεραρχία των πιστωτών ε, και της χαμηλής εξασφάλισης, της subordination. Ίσως με το ε, TILAC θα μπορούσαμε με το πιο, το, το πιο ουδέτερο ε, να εφαρμόσουμε αυτό το πρότυπο. Ίσως μπορεί να είναι η καλή προσέγγιση, η χρηματοπιστωτική κρίση πρέπει να μας οδηγήσει σε μακροοικονομική επίσης ε, προσέγγιση, αλλά όχι μόνο σε ε, μικροπροληπτική. Πιστεύω ότι στον ε, τομέα των τραπεζικό τα περισσότερα προβλήματα είναι μακροπροβλήματα και μια αυστηρή ε, προσέγγιση θα αυξήσει τα έξοδα των ε, τραπεζών, τα χρηματοπιστωτικά και θα μεταφερθούν ε, στους φορολογόμενους. Θα προτιμούσα να αυξήσουμε τις κοινέ μετοχές της κατηγορίας 1. Αυτό το μέσο να χρησιμοποιηθεί. Ίσως ε, η κεφάλαιο αυτό των κοινών μετοχών κατηγορίας 1, ίσως καλύτερη αναλογικότητα ε, για τις ε, μικρές. Δεν ξέρω πόσο, πόσα αποθέματα ασφαλείας θα έχουν οι τράπεζες και πότε θα έχουν επαρκή αποθέματα ασφαλείας. Είναι πρόβλημα της Κομισιό και Νομίζω ότι ε, εδώ ευνοείται η συμβατική ε, προσέγγιση για την απέτηση χαμηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας. Ε, τι περιστάσεις, οι πρόσφατες οι περιπτώσεις μας δείχνουν ότι θα προτιμούσαμε μια λύση όπου όλα τα μέσα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ε, πολύ γρήγορα για να μην έχουμε την αρχή περί επιδίνωσης της θέσης των πιστωτών. Υπάρχει λοιπόν ένα χάσμα το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί. Θέλουμε μια προσέγγιση πιο απλοποιημένη ότι όσο το δυνατόν νωρίτερα, τόσο καλύτερα να έχουν αυτά τα μέσα οι τράπεζες και θα θέλαμε μια ε, γεραρχία όπου όλα τα μέσα ε, να μπορούν να είναι ε, να λαμβάνονται υπόψη στην διάσωση με κάποια σειρά προτεραιότητας και αυτό είναι νομίζω μια προτεραιότητα και σχετικά με την οδηγία ανάκαψης και εξυγίανσης των τραπεζών. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, κύριο Σούρτας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λογική Σουρτάσον. Ευχαριστώ και τους κυρίους Χόκμαρ, ε, αλλά και τον κύριο Κάρας που παρουσίασε την εκθέση επί της ουσίας. Συμφωνώ με τους πράσινους όσον αφορά το άρθρο 20. Και εμεί θεωρούμε ότι η επαληφή αυτή τη αιτήσια προθεσμία δεν είναι καλή ιδέα γιατί ε, για τη διαχείριση του ρευστού είναι πάρα πολύ σημαντική η ρύθμιση. Έτσι, περιορίζουμε την αποτελεσματικότητα των TLIC. Αυτό που ακριβώς θέλουμε να αποφύγουμε. Οπότε και γι' αυτό θα, θα πρέπει να αναθεωρηθεί η ιδέα. Επίσης, όπως και οι πράσινοι και εμείς, θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να προλάβουμε και οι επαγγελματίες επενδυτές να μην χρησιμοποιήσουν αυτήν την ε, ρήτρα για το bail Και να δούμε τι θα γίνει με το MIFID και τα στοιχεία ενεργητικού που θα καλυφθούν. Μήπως αν ε, προβλέπετε ένα ελάχιστο επίπεδο επένδυσης τότε οι μη επαγγελματίες επενδυτέ να μην μπουν σε αυτή τη λογική, μην κάνουν τέτοια κίνηση. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Ευχαριστούμε εμείς, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Βάλλη. Ευχαριστούμε. Συμφωνώ με τον κύριο Τάσον. Θα πρέπει να υπάρχει μια προστασία όσον αφορά τα μέτρα που αφορούν το μπέιλιν για να προστατεύσουμε τους μικροκαταθέτες. Αυτοί δηλαδή που θέλουν να στραφούν προς τέτοια προϊόντα, δηλαδή για κάποια προϊόντα ασφαλιστικά, ε, ενεδρεύει κάποιος κίνδυνος. Οπότε μπορεί να πληγούν οι μικροκαταθέτες, οι πιο αδύναμες κοινωνικές τάξεις. Άρα εδώ θα έχουμε κάποια τροπολογία για το σημείο αυτό. Αυτό είναι το βασικό θέμα του οποίου προβληματιζόμαστε. Μάρκο Τζάνι, ευχαριστώ τον εισηγητή. Κάποια σημεία μας κάνουν να προβληματιστούμε. Είναι σημαντικά σε τη δική μας προσέγγιση αυτή την, την διαγραφή με την ετήσια προθεσμία και μας μας απασχολεί επίσης. Πρώτα πρώτα θα πρέπει να αποφύγουμε να υπάρχει αυτή η αναδρομική εφαρμογή των μέτρων κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με κάποιες εθνικές νομοθεσίες. Επίσης, θα πρέπει σε σχέση με, το, με την BRD BBRD, να δούμε τι θα γίνει με εκείνους οι οποίοι έχουν κάποιες μείζονες υποχρεώσεις. Γιατί αυτό φέρνει για τον Μπέιλιν αναδρομικότητα που δεν βοηθά τη διάσωση των τραπεζών. Οπότε είπαμε ότι αφού θέλουμε κάποια μέτρα προστασίας, αφού θέλουμε ένα μαξιλαράκι θα πρέπει να εξαιρέσουμε κάποια συγκεκριμένα ε, μέσα χρεωστικά. Τώρα, άλλα προβληματικά σημεία. Όσον αφορά την ευρύτητα και την ρευστότητα της αγοράς, όσον αφορά αυτά, τα στοιχεία, αυτή την κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, η εμπειρία μας λέει ότι όταν έχουμε όπως σήμερα τόσο μικρές αποδόσεις, οι θεσμικοί επενδυτές ενδιαφέρονται πάρα πολύ, είναι πολύ διαθέσιμοι να επενδύσουν αλλά για κάποια μέσα που προσφέρουν και προσφέρονται για υψηλές αποδόσεις. Το θέμα είναι βέβαια με ποιο κόστος και ποια θα είναι οι επιπτώσεις για τις τράπεζες, για τα συστήματα, τα τραπεζικά των χωρών που είναι πιο στριμωγμένες. Γιατί είδαμε ότι τα προβλήματα των τραπεζών ε, μεταφέρονται στην πραγματική οικονομία και κατόπιν στους καταναλωτές. Άρα θα πρέπει να εξεταστεί στην πραγματική οικονομία αυτά τα μέσα τι επενδύσεις θα έχουν. Αυτό, αυτό που είπαν οι δύο προηγούμενοι συνάδελφοι όσον αφορά την διαφάνεια, όσον αφορά την πώληση στην αγορά λιανικής για αυτά τα καινούργια ε, μέσα, για αυτού του είδους τα προνομιούχα, ομόλογα κλπ. Θα πρέπει να προσέξουμε και την διατύπωση. Θα πρέπει να μην ε, παρασύρεται ο επένδυτης για να αγοράσει αυτά τα μέσα. αυτά τα, την καινούργια asset class, αυτή την κατηγορία μέσων. Η Κεντρική Τράπεζα πριν από λίγες μέρες προειδοποίησε για τα προβλήματα ρευστότητας στις αγορές ομολόγων. Αληφθεί αυτό υπόψη και αυτά τα σημεία μας υπασχολούν και θέλουμε να τα συζητήσουμε με τον εισηγητή. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Μπορώ λοιπόν να δώσω το λόγο πάλι στον κύριο Κάρας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω στο όνομα του κυρίου Κούναρ Χόικμαρκ για τη συζήτηση αυτή. Θα αντιλαμβάνεστε ότι θα του μεταφέρουμε τις παρεμβάσεις σας και εγώ και η βοηθοί του που είναι παρόντες. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη συντομευμένη διαδικασία fast track. Στη διαδικασία αυτή δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αναλυτικές συζητήσεις όπως για άλλα θέματα. Όσον αφορά τις τροπολογίες 20 και 23 που αναφέρθηκαν, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο κύριος Χεκμαρκ έχει συμπεριλάβει εδώ προτάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και οι τροπολογίες αυτές αντιστοιχούν και στη δημόσια συζήτηση που έχει γίνει για το θέμα αυτό. Ο Σεπτέμβριος είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και ελπίζουμε έτσι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Εγώ ως κοιόδης της έκθεσης Σίμων θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια σειρά επικαλύψεων τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. όπως ε, για παράδειγμα στην οδηγία CAR και το άρθρο 52B. Ανασφάλεια των επενδυτών μπορεί να οδηγήσει και σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και δυσκολεύει και τη ζωή των οργανισμών. Γι' αυτό επικροτώ την πρόταση αυτή που επιφέρει περισσότερη ασφάλεια δικαίου. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστούν και τα κριτήρια υπολογισμού ε, των ε, MRL, των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, και να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη στο σύστημα. Νομίζω ότι έχει βρεθεί πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των κρατών μελών που ήδη έχουν αναλάβει σχετικά μέτρα Ε, και των άλλων και ο κύριος Χεκμαρκ όπως και ο κύριος Σίμων θα επιδιώξουν ευρεία πλειοψηφία και ευρεία συνένεση στις επόμενες τροπολογίες. Καλό είναι λοιπόν να αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. I would like... Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω αυτό που είπε ο κύριος Κάρας ε, στο όνομα του εισηγητή. Ε, είναι διαδικασία συντομευμένη, ισχύει το άρθρο 108 του κανονισμού. Είναι με ευπρόσδεκτες ή τροπολογίες για το θέμα αυτό, όχι όμως για το υπόλοιπο, για το βασικό πακέτο ε, και θα θεωρηθούν απαράδεκτες τέτοιες τροπολογίες. οι τροπολογίες λοιπόν θα πρέπει να αναφέρονται στο τμήμα Fast Track και το, οι υπόλοιπε τροπολογίες θα συζητηθούν εν ευθέτω χρόνο. Ναι, πράγματι, ξέρω ότι πρόκειται για άλλη πρόταση, αλλά ουσιαστικά ε, έχει να κάνει με το ίδιο θέμα. Μπορεί λοιπόν οι ευρωβουλευτές ε, να ε, το εκμεταλλευτούν ώστε να τροποποιήσουν άλλα πράγματα. Να επικεντρωθούμε λοιπόν στο άρθρο 108 και τη θέση σε ισχύ. Άλλε τροπολογίε ε, δεν θα θεωρηθούν παραδεκτέ. Το χρονοδιάγραμμα έχει ω εξή. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 4 Ενάτου, εξέτασή τους 25 Ενάτου, ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ 25 Σεπτεμβρίου και κατόπιν τριμερής διάλογη. Προτείνω 4 λεπτά διάλειμμα, προτού προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες όπως ε, προβλέπετε στις 12.30. Ευχαριστώ. Dear colleagues, may I ask you to take seat. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ζητώ να καθίστε, παρακαλώ. Να βάλετε την ε, κάρτα ψηφοφορίας ε, για να ψηφίσουμε. Ε, κάνουμε μια δοκιμή τώρα. keep it open. Wait, I, wait, I tell you. Please, colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ. Ποιος λείπει. Still one colleagues to vote, but still some... Κάποιοι ακόμα απουσιάζουν. Για να δούμε ποια είναι η πλήρη σύνθεσή μας. Giving the time if... Okay. Σας δίνω λίγο χρώμα ακόμα. Please. Colleagues, put... Παρακαλώ συνάδελφοι, τοποθετήστε την ε, κάρτα στη συσκευή. Ραμόν, you can also vote. Ραμόν, και εσύ μπορείς να ψηφίσεις, δοκιμή κάνουμε. Jezek also, so we are now 46, very good. Okay, the test is closed and we now will vote a number of uh, uh, provisional agreements. So... Έχουμε μια σειρά ε, προσωρινών συμφωνιών ε, για να ολοκληρώσουμε στην πρώτη ανάγνωση ε, κάποια θέματα. Συγχαίρω όλους τους εισηγητές και το πρώτο θέμα είναι οι κοινοί κανόνες για την τιτλοποίηση. Αρχή της ψηφοφορίας. No. Yes, it's roll call vote. Again, the vote is open again. Ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας εκ νέου. Processed as a roll call vote. Now we have to. Διότι δεν ήταν ονομαστική. still colleagues to vote if they wish. Παρακαλώ, αν επιθυμεί κανείς να ψηφίσει, προλαβαίνει. Α, επιτέλους ο εισηγητής υπερψήφισε την πρότασή του. Ωραία. understand colleagues do not wish to vote. Από ό,τι καταλαβαίνω, δύο συναδελφοί δεν θέλουν να ψηφίσουν, δικαίωμά τους, λήξη της ψηφοφορίας. 34 υπέρ, 12 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Επίκαιρο θέμα, όπως και το επόμενο, με εισηγητή τον Ότμαρ Κάρας. Πρόκειται για το άλλο τμήμα του STS, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας. Okay. We can close. Λήξη. 35 υπέρ, 12 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια και στον Ότμαρ Κάρας. Τώρα έχουμε στατιστικό θέμα. που είχε αναλάβει το ε, Προεδρείο, εισηγητή ο Πρόεδρο, ε, όπω δυστυχώ συχνά γίνεται, έναρξη τη ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Λήξη τη ψηφοφορία. 39 υπέρ, 3 ψήφοι κατά, 6 αποχέ. Σα ευχαριστώ. Προχωράμε στην έκθεση Πιέτη Κάινεν σχετικά με το, τα επιχειρηματικά κεφάλαια και το Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Έναρξη της ονομαστικής ψηφοφορίας. closed. Λήξη της ψηφοφορίας, 38 υπέρ, 2 κατά, 7 αποχές. Συγχαρητήρια και στη ΣΥΡΠΑ. Και προχωράμε τώρα στην έκθεση Πίτερ Ζήμων που μόλις συζητήσαμε με συντομευμένη διαδικασία σχετικά με το ΔΠΧ α9 και τα μεγάλα νύχματα. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Σ γάμα υπέρ κατά υπέρ είστε υποθέτω ε. ε το χέρι σας όμως όταν είπα κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική, ε, τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική D δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Όπως θα προσέξατε, κάποιες ε, τροπολογίες θεωρήθηκαν μη παραδεκτές ε, διότι ξεπερνούσαν το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας Fast Track. Θα μπορέσετε να υποβάλλετε τις τροπολογίες αυτές στο πλαίσιο του κανονικού πακέτου. Δίνουμε και λίγο χρόνο στην Έστερ Λάνια να ψηφίσει. Α, α, α, παράνομο ήταν αυτό. Τέλος πάντων, για καλό σκοπό γίνονται όλα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λήξη της ψηφοφορία. 39 υπέρ, 11 κατά. Καμία αποχή. Πρέπει να ψηφίσουμε κάποιες τροπολογίες στο νομοθετικό ψήφισμα. 26 υπέρ, κατά αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 30 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το νομοθετικό ψήφισμα θεωρείται ότι εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε την απόφαση για έναρξη των διοργανικών ε, διαπραγματεύσεων με ονομαστική ψηφοφορία. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας υπέρ 40, 11 κατά, 0 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν η απόφαση. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και στους σκιώτες. Okay, so we can close the meeting. Λήξη της συνεδρίασης. Θα συνεχίσουμε στις 4. Ευχαριστώ πολύ.